Nous allons commencer notre réunion. Ξεκινάμε. Παρακαλώ να καθίσετε. καλωσορίζω λοιπόν όλους. Συνοντόμεθα με αφορμή την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας το 2013. Σας εύχομαι λοιπόν καλή χρονιά σε όλους. Έχουμε πολλά θέματα μπροστά μας. Έχουμε το μέσο για την ανάπτυξη και τη συνεργασία, την δημιουργία του Εθελοντικού Ευρωπαϊκού Σώματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας, τους στόχους της χιλιετίας και την προετοιμασία του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου σχετικά με το ΦΕΝΤ και υπάρχουν και άλλα βέβαια και όχι μόνο τα αυτά που προείπα. Δύσκολα θέματα σε μια δύσκολη περίοδο και πολλοί εδώ θα θεωρούσαν σωστό να κάνουν δραστικές περικοπές στην προσπάθεια για την ανάπτυξη, το οποίο πολλοί λέγουν ότι έχει καταδικαστεί πλέον το πρόγραμμα για την ανάπτυξη οικονομικά. Εμείς είμαστε εδώ όμως για να διαψεύσουμε αυτές τις προφητείες. Πρέπει να εμείνουμε στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων στις οποίες θα πάρουμε μέρος και σε όλα τα φόρα στα οποία θα μιλήσουμε πρέπει οι απόψεις μας να ακουστούν. Είναι δύσκολο να μην συζητήσουμε επίσης και για την κατάσταση στο Μαλί. Πιστεύω, όπως και οι περισσότεροι συνάδελφοι, ότι η παρέμβαση αυτή στρατιωτική της Γαλλίας ήταν δικαιολογημένη, αλλά πρέπει να είναι περιορισμένη στο χρόνο και αφρικανικά στρατεύματα θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να αντικαταστήσουν τους Γάλλους στο Μαλί. Όμως ο πόλεμος αυτός είναι αποτυχία. Είναι αποτυχία λόγω δύο άλλων αποτυχιών, της πολιτικής αποτυχίας και της αποτυχίας της προσπάθειας να σωθεί το Μαλί από τη φτώχεια. Γιατί έχουμε πει εμείς ότι στην μη ανάπτυξη και στην μιζέρια ο ριζοσπαστικός ακραίος αυτός ακτιβισμός ο θρησκευτικός ριζώνει και δυστυχώς εμείς δεν μπορέσαμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και πολλές φορές και οι διαφορετικές παρεμβάσεις πολλές φορές προκάλεσαν χειρότερα προβλήματα από αυτά τα οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και πολλές φορές επιβάλλονται στις υποανάπτυξη χώρες παρά τις προσπάθειες που κάνουν. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε στο μέλλον μετά την παρέμβαση αυτή η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και η ε, δημιουργία ενός δημοκρατικού διαλόγου που λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των μειονοτήτων θα οδηγήσει σε μια δίκαιη ανάπτυξη, θα επιτρέψει τη διασφάλιση στην, ε, στα τρόφιμα και είναι όλα αυτά προϋπόθεση για μια διαρκή ειρήνη στο Μαλί. Άμεσα τώρα η ανθρωπιστική κατάσταση θα πρέπει να προκαλέσει την προσοχή μας. Μέχρι τώρα έχουν εκτοπιστεί 400.000 κάτοικοι. Η κρίση στον τομέα των τροφίμων φύγει 18 εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής που φεύγουν από τις επιθέσεις των τζιχαντιστών και από τις μάχες. Η κυρία Άστον έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η βοήθεια η ανθρωπιστική προς το Μαλή θα συνεχιστεί και θα αυξηθεί έτσι ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού. Είμαι πεπισμένη ότι η Επίτροπος Γεωργίευα όπως πάντα θα έρθει εδώ και θα αναφερθεί στην Επιτροπή μας για τους στόχους τους οποίους έχει και να μας δώσει τις πληροφορίες που έχει. Τώρα λοιπόν περνάμε στο κανονικό κομμάτι. Υπάρχει μια μικρή τροποποίηση. Η κυρία Λούλινγκ πρέπει να είναι παρούσα στην ε, Επιτροπή Αλληλεία σήμερα το απόγευμα και έτσι η παρουσίαση της νομοδότησής για τη συμφωνία την Αλληλευτική με την Μάδα Αγασκάρη θα είναι το τελευταίο θέμα για σήμερα. Λοιπόν, έγινε η μικρή αυτή τροποποίηση στην μερισία διάταξη. Λάβατε και τα πρακτικά της συνεδρίασης της 6 Δεκεμβρίου του 12. Αν έχετε παρατηρήσει σχετικά με τα πρακτικά αυτά, θα πρέπει να τις διατυπώσετε στη γραμματεία πριν από το τέλος της συνεδρίασής μας, γιατί ε, διαφορετικά τα πρακτικά αυτά θα θεωρηθούν δεκτά λάβατε τις συστάσεις και τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης των συντονιστών της 13ης και 18ης Δεκεμβρίου του 12. Αν έχετε παρατηρήσει σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, να τα μεταφέρετε στη γραμματεία πριν από το τέλος της συνεδρίασης, άλλως ε, τα, ε, ε, τα αποτελέσματα αυτά θα γίνουν δεκτά. Τώρα πρέπει να σας κάνω και μια ανακοίνωση. Προεδρεύω μαζί με τον κύριο Μπροκ της Επιτροπής Εκλογικής Παρατήρησης, Εκλογικής Εποπτείας και γι' αυτό θα ήθελα να κάνω τις εξής συστάσεις, λέει η κυρία Ζολή. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε αιτήσια βάση σε αποστολές παρατήρησης εκλογών που έχουν σαν στόχο την ενίσχυση της εκλογικής διαδικασίας και της νομιμότητας της διαδικασίας αυτής σε εθνικό επίπεδο, το ότι η διεξαγωγή των διαδικασιών των εκλογικών να είναι η πιο σωστή και διαφανής που μπορεί να γίνει. Αυτό είναι απαραίτητη δημοκρατική προϋπόθεση για την ανάπτυξη κάθε χώρας. Υπάρχει λοιπόν ο στόχος της καλύτερης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνεισφορά στην επίλυση των διαφορών και τη σταθεροποίηση των κρατικών δομών μετά το τέλος των εχθροπραξιών. Οι ε, αποστολές αυτές διεξάγονται κυρίως στις χώρες ΑΚΕ και τα μέλη της Επιτροπής μας έχουν όχι μόνο όλες τις ε, γνώσεις που χρειάζεται, αλλά έχουν και ίδιο ενδιαφέρον θα έλεγα για τα θέματα και γι' αυτό στην τελευταία επιστολή την οποία ε, στείλαμε με τον κύριο Μπροξ την κυρία Άστον, τη ζήτησα να σεβαστεί μια κάποια ισορροπία ανάμεσα στην Επιτροπή μας και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στον ορισμό των αρχηγών των αποστολών αυτών εκλογικής παρατήρησης. Σας ενθαρρύνω λοιπόν όλους να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες της ομάδας στήριξης της δημοκρατίας και συντονισμού των εκλογών, να συμμετέχετε σε τέτοιου είδους αποστολές, κυρίως εφόσον δεν το έχετε κάνει, και θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τους συναδέλφους της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και έτσι θα μπορέσετε να γίνετε υπεύθυνοι των αποστολών αυτών και εσείς όπως και αυτοί. και να μεταφέρετε μετά το τέλος της αποστολής σας, της παρατηρήσεις σας στην Επιτροπή μας. Λοιπόν, το λόγο τώρα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πιθανές παρατηρήσεις αυτά τα οποία σας είπα. Ευχαριστώ. Λέγομαι Πίτε Κρέγκλ. Από τον Νοέμβριο είμαι υπεύθυνο για τα διοργανικά θέματα και τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν συνεργαζόμαστε με το Κοινοβούλιο και τους, τα, θεσμικά όργανα με τις συνδεδεμένες χώρες. Θα ήθελα να σας αναφέρω ορισμένες από τις επερχόμενες πρωτοβουλίες της Κομισιόν για το επόμενο εξάμενο, κάποιες από τις οποίες γνωρίζετε. Ένα σημείο το οποίο θα συζητηθεί αύριο στην ακρόαση για τους ε, στόχους της χιλιετίας, τους στόχους της χιλιετίας. Ήθελα να επιβεβαιώσω ότι έχουμε μία ανακοίνωση που πρόκειται να υιοθετηθεί τέλη Φεβρουαρίου με τίτλο παρακολούθηση της στρατηγικής ε, των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας για την προετοιμασία της συνεδρίασης στη Νέα Υόρκη το φθινόπωρο φέτος ε, προετοιμασία του πλαισίου μετά το 2015 και την παρακολούθηση της ε, σύσκεψης Ρίο συν Ετοιμάζεται λοιπόν αυτή η ανακοίνωση από κοινού υπό τους επιτρόπους Πίμπαλτς και Ποτότσνικ για τα θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Επίση, θα σα αναφέρω κάποιε ανακοινώσει ε, για τα θέματα τη διατροφή και τη διατροφική ασφάλεια, όπου έχουμε πρώτα απ' όλα ένα σχέδιο υλοποίηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για αρρωγή προ αναπτυσσόμενε χώρε για αντιμετώπιση των προκλήσεων διατροφή που πιστεύω ανέφερε ο κ. Πίμπαλξ το Δεκέμβριο ενώπιον τη Επιτροπή σα. Δεύτερον, μια ανακοίνωση για την διατροφή ε, για μητέρες και βρέφη και τρίτον μια εκθέση για την ε, διατροφική διευκόλυνση, δηλαδή διευκόλυνση για ταχεία απόκριση για την αντιμετώπιση των τιμών, των θεμάτων τιμών σε αναπτυσσόμενες χώρες. Το πρώτο που αφορά τη διατροφική ασφάλεια και τις σχετικές προκλήσεις ε, θα βοηθήσει να επιταχύνουμε την καταπολέμηση της έλλειψης διατροφής και την ανάπτυξη ενός ε, επιχειρησιακού πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ενισχυθεί ο συντονισμός και η λογοδοσία των δράσεών μας. Το δεύτερο που αφορά τη διατροφή για μητέρες και βρέφη και τη σχετική έρωγη, οφείλεται στο γεγονός ότι δεσμευόμαστε όλο και περισσότερο στην καταπολέμηση της ε, ελλειπούς διατροφής. Πρέπει να διασφαλίσουμε συνοχή πολιτικών μεταξύ αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών ε, προοπτικών όσον αφορά τη διατροφή, αλλά και μεταξύ των πολιτικών κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το τομέα. Και τρίτον θα υπάρξει μια εκθέση για την υλοποίηση του Food Facility, της διευκόνησης για τη διατροφή σε διάστημα τριών ετών που αναμένει θετική απόκριση από τις χώρες και περιφέρειες στόχους, μετριάζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις των τιμών των τροφίμων στους σχετικούς πληθυσμούς και αυξάνοντας ε, τις ικανότητες και τη διακυβέρνηση στις χώρες αυτές. Η ανακοίνωση και τα σχετικά έγγραφα θα εξετάζουν τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονται και τα διδάγματα που έχουν αποκομιστεί. Μιλάμε λοιπόν για ένα πακέτο τριών σχετικών εγγράφων για τη διατροφική ασφαλεία και τη διατροφή. Φυσικά υπάρχουν και άλλα σημεία στο πρόγραμμα εργασία μα, αλλά πιστεύω έχετε ήδη εξοικειωθεί με αυτά. Αυτά είχα να σα πω προ το παρόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν έχουμε λάβει ερωτήσεις ε, προς την Επιτροπή. Θα περάσουμε λοιπόν αμέσως στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης που έχει ένα διπλό στόχο την απαλλαγή 2011 για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τμήμα 3 και επίσης την απαλλαγή 2011 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Τέις Μπέρμαν, στον οποίο δίνω τον λόγο αμέσως. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα λοιπόν τα Ολλανδικά και για την χορήγηση απαλλαγής για το Αναπτυξιακό Ταμείο σε σχέση με αυτό ίσως εκ προημίου μια παρατήρηση. Δεν αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα όταν πρόκειται για χορήγηση απαλλαγής γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει τα κείμενα βέβαια. Πρέπει αποκλειστικά να βασιζόμαστε σε στοιχεία και δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελεκτικού Συνεδρίου. Και είναι αυτονόητο ότι εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο του ελεγκτικού συνεδρίου και είναι αυτονόητο ότι κατανοώ και τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την πλευρά της. Όμως είμαι κάπως αμήχανος διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί ανεξάρτητα το ίδιο να εξετάσει αυτά τα οποία διαπιστώνει ή διαπίστωσε το ελεγκτικό συνέδριο ή τι έγινε επιτόπου όσον αφορά τα τελικά συμπεράσματα που συντάσσει και διατυπώνει το ελεγκτικό συνέδριο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια παραδείγματα για τέτοιες περιπτώσεις. Μπορεί να διατυπώνει κανείς ερωτήματα, για παράδειγμα, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ευρωκοινοβούλιο έχει και εκείνο τρεις ε, στόχους, νομοθετικό έργο, η απήχηση των απόψεων και των ε, ε, θέσεων των πολιτών της Ευρώπης και η άσκηση ελέγχου. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό, τον έλεγχο, σε σχέση με την πολιτική, καμιά φορά δεν πράμε πολύ καλά, δεν έχουμε πολύ καλές επιδόσεις. Είμαστε αδύναμοι σε αυτό το πεδίο, θα έλεγα. Το κατανοώ οπωσδήποτε από την άλλη πλευρά, ότι εμείς την πολιτική, ας το πω έτσι, από πλευράς πολιτικής δεν είναι εύκολο να ελέγχει κανείς απόλυτα. Έχουμε όμως και τις παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου που προστίθενται σε, αυτές τις, σε αυτή την κατάσταση και στη χορήγηση απαλλαγής για το Αναπτυξιακό Ταμείο διαπιστώνει κανείς ένα συγκεκριμένο ποσοστό σφάλματος 5,1% το 2011 παραπάνω δηλαδή από το 2010 που ήταν 3,4% τότε. Τίθεται το ερώτημα από πού προέρχεται αυτή η κατάσταση, σε τι οφείλεται το σύστημα ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα τεκτενόμενα του Αναπτυξιακού Ταμείου εν μέρη αποτελεσματικό θεωρείται από το ελεγκτικό συνέδριο. Εν μέρη θετικό, εν μέρη όμως ε, και μη αποτελεσματικό. Υπάρχουν κενά σε σχέση με τον έλεγχο φαίνεται. Και αυτό συναρτάται από το ότι οι αντιπροσωπείες μας σε σχέση με διάφορε χώρε δεν έχουν αρκετά στελέχη και δυσχεραίνεται το έργο του. Σε κάποιε απαντήσει, λέει το η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το κείμενο του ελεγκτικού συνεδρίου ότι έχουν προσεγγιστεί όλα αυτά με τέτοιο τρόπο ώστε λιγότερα στελέχη θα είναι καλύτερα καταρτισμένα με καλύτερε, με καλέ υψηλέ επιδόσει. Πράγμα που σίγουρα δεν είναι καθόλου απλό φοβούμε. Καθόλου απλό αυτό το έργο και αδειμονώ μήπω θα μπορούσε να συμπληρώσει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτέ τι τοποθετήσει τη με λιγότερα στελέχη να υπάρχει μεγαλύτερη πραγματογνωμοσύνη και αποτελεσματικότητα Ίσως αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί, διότι σε σχέση με τι διαπραγματεύσει ε, για τα πολιετή προγράμματα, ίσω θα μπορούσε κάτι να πορεύσει εκεί. Θα ήταν ενδιαφέρον ίσω. Διαπιστώνεται λοιπόν με δειγματοληπτικούς ελέγχους που γίνονται σε σχέση με τις πληρωμές, πληρωμές δηλαδή για παράδειγμα διεθνών ε, οργανισμών. Ερώτηση προς την Επιτροπή. Αυτό το ποσοστό σφάλματος μπορεί να οφείλεται σε κάποια συγκεκριμένα αίτια που θα μπορούσαν ίσως να αντιμετωπιστούν και να καταπολεμηθούν. 50% των πληρωμών έχουν κάποιες παρατυπίες ή κάποια προβλήματα. Ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια αποτελεσματικότητα μπορεί να αναμένει κανείς με λιγότερα στελέχη και μεγαλύτερη πραγματογνωμοσύνη ποια αποτελέσματα μπορεί να έχει κανείς και μία τοποθέτηση σε σχέση με την εκτέλεση των προγραμμάτων όσον αφορά τις υποδομές αυτού του είδους ε, τα θέματα ε, έμειναν πολύ πίσω από τους στόχους ε, σε μεγάλο ποσοστό πίσω από τον στόχο του 2011. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι πράττει για να βελτιωθούν τα πράγματα και να αλλάξει αυτή η κατάσταση πράγματων για τη χορήγηση απαλλαγή και για την απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να συνεχίσω, Πρόεδρε, με αυτό το θέμα για την απαλλαγή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, εντάξει, πολύ καλά. Λοιπόν, καλύτερα φαίνονται τα πράγματα σε σχέση με αυτό. Εξωτερική βοήθεια, ευρωπαϊκή προϋπολογισμός σε αντίθεση με τον προϋπολογισμό του Αναπτυξιακού Ταμείου για παράδειγμα. Εκεί έχουμε ένα ποσοστό σφάλματος που βρίσκεται κάτω από την θα έλεγε κανείς ε, στατιστική ε, σπουδαιότητα, κάτω δηλαδή από το ποσοστό σφάλματος το οποίο θα μπορούσε να θεωρείται ε, συστημικά δεδομένο. Ωστόσο, με τους ελέγχους τα πράγματα δεν βελτιώνονται υποχρεωτικά όταν έχουμε χρήση ε, στελεχών ε, σε σχέση με, για παράδειγμα, την διπλωματική υπηρεσία. Παράδειγμα, το 2011, 43 άτομα χρησιμοποιήθηκαν για τέτοιου είδους ε, καθήκοντα. Γνωρίζουμε βέβαια ότι μπορούν να μετατίθενται τέτοιου είδους υπάλληλοι, αλλά αυτό ξεπερνά το πλαίσιο της ελαστικότητας ή ευελιξία 43 στελέχη. Καλό θα ήταν αν η διπλωματική υπηρεσία θα μπορούσε να σεβότανε τις ε, συμφωνίες και τα όσα θα έπρεπε να ισχύουν ε, με την εξωτερική βοήθεια διότι δεν, δεν υπάρχουν τα στελέχη ούτως ή άλλως. Οι υπάλληλοι δεν υπάρχουν και στο τέλος τέλος έχουμε μετρήσιμους δείκτες. Μετρήσιμοι δείκτες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων. Θα πρέπει γοργά να εισαχθούν αυτοί οι δείκτες, ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε μια ε, διευκόλυνση και ελάφρυνση, ανακούφιση του προσωπικού Αυτά είχα να πω, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ε. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στην Επιτροπή. Η Γενική Διεύθυνση ΔΕΒΚΟ, κύριε Σαμέλ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που μας δίνεται η ευκαιρία να σας εξηγήσουμε λίγο τι γίνεται στην Επιτροπή τι βλέπουμε να παρουσιάζεται ως πρόβλημα το 2012. Θα αναφερθώ στα ερωτήματα του εισηγητή και θα προσπαθήσω να τα απαντήσω ένα προς ένα για να είναι πιο απλή η συζήτηση. Ξεκινάμε λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το 5,1% σφάλματος, ποσοστό σφάλματος. Υπάρχουν δύο τρόποι να το δούμε αυτό το ποσοστό σφάλματος, είτε αύξηση τα δύο τελευταία χρόνια, είτε σταθεροποίηση τα τελευταία δέκα χρόνια. Διότι το ελεκτικό συνέδριο μας είπε ότι από το 2007, από το οποίο ξεκίνησε να μας δίνει στοιχεία, το ποσοστό σφάλματος ήταν μεταξύ 2 και 5% εκτός από πριν δύο χρόνια όπου ήταν χαμηλότερο και φέτος όπου είναι 5,1%. Δηλαδή υπερβαίνει το ανώτατο όριο κατά 0,1%. Αυτό το στοιχείο το 5,1 φυσικά το αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα, διότι θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Μπορώ να σας πω εγώ λοιπόν τι κάναμε αμέσως μόλις ε, αντιληφθήκαμε αυτό το ποσοστό σφάλματος. Το πρώτο που κάναμε ήταν ότι διαπιστώσαμε πως αυτό το ποσοστό σφάλματος ε, προερχόταν από δύο αντιπροσωπείες είναι τυχαίο όπως είπε το, είναι το, η τυχαιότητα των δειγματοληψιών όπως είπε ο υπεύθυνο του ελεκτικού συνεδρίου. Στείλαμε μια αποστολή για να ελέγξει το σύστημα ελέγχου αυτών των δύο αντιπροσωπιών και ένα σχέδιο δράσης προτάθηκε αμέσως στην Κομισιόν, στην έδρα. Ελπίζουμε ότι θα δούμε τα αποτελέσματα μέσα στο 2013. Για να απαντήσω τώρα σε μια άλλη ερώτηση από τότε, αυτό που κάναμε ήταν αυτό που λέμε εκ νέου ανάπτυξη. Εξετάσαμε τις ανάγκες σε όλες τις αντιπροσωπείες. Είναι τεράστια η εργασία, είναι η πιο μεγάλη επανάληψη ανάπτυξη, ας πούμε, επανεξέταση ουσιαστικά του deployment. Παρατηρήσαμε έλλειψη ε, διαπιστευμένου προσωπικού, πιστοποιημένου προσωπικού, εξειδικευμένου προσωπικού, ειδικά στην Αφρική και στην Λατινική Αμερική και στην Ασία όπου υπάρχουν πολλές αναδυόμενες χώρες που δεν έχουν πια τα προβλήματα που είχαν κάποτε και μετατοπίζεται στο προσωπικό προς την Αφρική ένα άλλο στοιχείο η Αφρική, την Αφρική και οι γειτονικέ της χώρες ε. ένα άλλο σημείο ότι αυτή τη στιγμή εξετάζονται όλες οι ικανότητες εντός των αντιπροσωπείων και στην έδρα ώστε να εντοπίσουμε της ελλείψεις ικανοτήτων ή της ελλείψεις ε, ατόμων επαρκώς εξειδικευμένων σε σχέση με τα μολυντικά προγράμματα που θα αποφασιστούν. Έτσι θα μπορέσουμε να ανακατανύμουμε το ανθρώπινο δυναμικό ανάλογα με τις ανάγκες. Εξάλλου γνωρίζετε ότι προτάθηκε να κάνουμε αυτό που ονομάζουμε σε άπτες τα ελληνικά hubs, κόμβους δηλαδή, όπου θα συγκεντρώνουμε ε, έμπειρους ανθρώπους, ε, ειδικότερα σε δημοσιονομικά θέματα. Έτσι ελπίζουμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα των ε, έμπειρων ειδικών. Ένα άλλο σημείο, η ΔΕΒΚΟ, με το Γενικό της Διευθυντή, αποφάσισε να διαιρέσει το τμήμα Αφρικής σε δύο διευθύνσεις. Το Αφρική 1 που προλαμβάνει την Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική και το 2, το δεύτερο τμήμα που, που περιλαμβάνει τη Δυτική και την Υποσαχάρη Αφρική. Έτσι ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλύτερη παρουσία και ο διευθυντή ε, θα ενημερώνεται καλύτερα για το τι συμβαίνει στην κάθε αντιπροσωπεία, θα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα διάφορα προβλήματα σε θέματα ελέγχου. Τέλος, ε, αποφασίστηκε από το 2011 να ζητάμε από τους επικεφαλείς αντιπροσωπιών να υπογράφουν ένα statement of assurance, όπως λέμε στα αγγλικά, δήλωση διασφάλισης, ώστε να αναφέρουν καλύτερα το ελεγκτικό τους έργο στις αντιπροσωπείες τους. Αυτή η διασφάλιση, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι, θα επιτρέπει στους γεωγραφικούς και θεματικούς διευθυντές να συμβάλλουν πολύ πιο ουσιαστικά στην ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή Φυσικά αυτό το σύστημα ξεκίνησε το 2011, όπως όλα τα συστήματα είναι σχετικά καινούριο και έχει κάποια ελαττώματα σε αυτές τις πρώτες φάσεις. Έχουμε διάφορα προβλήματα με τους δείκτες, αλλά στους δείκτες θα επανέλθω, γιατί δεν κατάλαβα πολύ καλά για ποιους δείκτες μιλήσατε κύριε Μπερμαν, αλλά έχουμε κάποιους εδώ δείκτες κλειδιά προγραμματισμού που χρειάζονται αναθεώρηση ή προσαρμογή, ώστε να είναι καταλληλότεροι τελευταίο σημείο. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή εξετάζει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην έκθεσή του ώστε να οργανώσει αποστολές ε, στις διάφορες χώρες ε, για τα ίδια τα έργα και αποστολές ε, που θα περιλαμβάνουν μέλη ομάδων οικονομικού ελέγχου, ελέγχου και οικονομικών αυτή τη στιγμή μελετάμε την πτυχή κόστους αποτελεσματικότητας. Γίνονται διάφοροι έλεγχοι. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην καταλήξουμε σε κάτι αναποτελεσματικό. Αυτά είχα να σας πω όσον αφορά την αντίδρασή μας στο 5,1% του ΕΤΑ. Να περάσουμε τώρα στους διεθνείς οργανισμούς. Μας ενδιαφέρει αυτό το πρόβλημα. Έχουμε δύο μείζωνα προβλήματα το πρώτο ήταν διαφορά ερμηνεία μεταξύ τη Κομισιόν και των διεθνών οργανισμών όσον αφορά τι ενισχύσει, τη πληρωμή που βασίζεται στο γνωστό ΦΑΦΑ. Αυτό το έχουμε ρυθμίσει και οι δαπάνε θα καταβάλλονται εφόσον έχουν ε, πραγματοποιηθεί υλοποιήσει και όχι δεσμεύσει των διεθνών οργανισμών. Αυτό το λύσαμε λοιπόν φέτο το 2012 και ελπίζω ότι αυτό το είδο ποσοτικοποιημένου σφάλματο θα εξαφανιστεί. Επιπλέον, όσον αφορά τα 18 λάθη που εντόψε το Ελεκτικό συνέδριο για του διεθνεί Οργανισμού, τα 12 αφορούν την Μισόμ, δηλαδή την αποστολή στη Σομαλία. Αμφισβήτησε η Κομισιόν αυτά τα σφάλματα για δύο λόγους. Το ελεκτικό συνέδριο θεώρησε ότι υπήρχε κίνδυνος διπλής πληρωμής των στρατιωτών. Εμείς επικοινωνήσαμε με τους άλλους οργανισμούς, τους κυριότερους κυρίως της, ε, τα Ηνωμένα Έθνη, και τον Αφρικανικό Οργανισμό και το USA και αντιληφθήκαμε ότι το USAID και τα Ηνωμένα Έθνη δεν πλήρωναν τους στρατιώτες. Ουσιαστικά ο κίνδυνος ήταν ελάχιστον. Επαληθεύσαμε, ζητήσαμε έναν έλεγχο για να επαληθεύσουμε ότι στο 2012 δεν γινόταν αυτές οι πληρωμές. Ο κίνδυνος ήταν εξαιρετικά χαμηλός, είναι εξαιρετικά χαμηλός και πιστεύουμε ότι αυτός ο κίνδυνος που εντόπισε το ελεκτικό συνεδρίο, χωρίς να τον ποσοτικοποιεί, κατά την άποψή μας είναι ανύπαρκτος. Το δεύτερο σφάλμα που εντόπισε το ελεγκτικό συνέδριο επισημαίνει ότι η Κομισιόν δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει κατά πόσο πληρώθηκαν οι ίδιοι στρατιώτες. Η Κομισιόν ανέθεσε αυτό το καθήκον στην Αφρικανική Ένωση με εκθέσεις της Αφρικανικής Ένωσης που μας ε, επιτρέπουν να δούμε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Μετά από αυτή την παρατήρηση του ελεκτικού συνεδρίου ζητήσαμε έκθεση ακόμα πιο ακριβή και οικονομικό έλεγχο ακόμα πιο ενδελεχή ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι στρατιώτες λαμβάνουν τις αμοιβέ τους. Δεν είχαμε καμία, ε, ε, κανένα αίτημα από τα υπηρετούντες. Λοιπόν, αυτός ο κίνδυνος θα υπάρχει πάντα διότι η Κομισιόν δεν είναι αυτή που πληρώνει τη μισθοδοσία των στρατιωτών. Δεν έχουμε τέτοια μέσα. Εάν λοιπόν αφαιρέσουμε αυτά τα 12 ασφάλματα, 2 επί 6 δηλαδή της μη σώμα, τα 3 ασφάλματα που έχουν ήδη διορθώθει, θα δείτε ότι το ζήτημα των διεθνών οργανισμών μειώνονται από 18 σε 3. Τρία μικρά προβλήματα που αυτή τη στιγμή εξετάζουμε είναι ad hoc προβλήματα, ουσιαστικά μετάδοση πληροφοριών, έγκαιρη μετάδοση των πληροφοριών και παρόμοια. Ελπίζω λοιπόν ότι θα ξεφουσκώσει το ζήτημα αυτό που τέθηκε με τη Μισόμ. Τώρα όσον αφορά το πρόβλημα προσωπικού, όπως σας είπα προηγουμένως, ε, ανακατανέμουμε το προσωπικό προς την αντιπροσωπεί με τις μεγαλύτερες ανάγκες. Δηλαδή έχουμε λιγότερο προσωπικό, το οποίο όμως ε, αποστέλλεται εκεί όπου είναι αναγκαίο και φροντίζουμε οι έμπειροι, τα έμπειρα άτομα να βρίσκονται εκεί όπου χρειάζονται. Δεν θα γίνει αμέσως, θα χρειαστούν 2-3 χρόνια. Ελπίζουμε ότι το 2014 όταν ε, θα γίνει ο νέος προγραμματισμός θα έχουμε επαρκές προσωπικό εκεί όπου είναι αναγκαίο και στα hubs, στους κόμβους αυτούς. Συνεχίζουμε την κατάρτιση του προσωπικού. Θεωρούμε ότι υπάρχει ήδη τεράστια κατάρτιση, αλλά υπάρχει μεγάλη εναλλαγή προσωπικού, ειδικά με του συμβασιούχου. Χρειάζονται κατάρτιση όσον αφορά του ελέγχου. Θεωρούμε ότι υπάρχει ένα σημείο που θα έπρεπε να ενισχύσουμε την κατάρτιση και το μελετάμε αυτή τη στιγμή. Αφορά τι προσκλήσει για υποβολή προσφορών, όπου παρατηρήσαμε κάποιο μικρό πρόβλημα. Το τελευταίο σημείο που αφορά το ΕΤΑ είναι το πρόγραμμα υποδομών. Οι καθυστερήσεις σε γενικές γραμμές αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά είναι τεράστιες υποδομές γενικά, οδοί, ε, παροχή νερού ε, και έχουμε άλλο ένα πρόβλημα της εγγύησης ε, για να διασφαλιστούν αυτές οι εργασίες και αυτές οι εγγύσεις δεν παρέχονται από, τους, από όσους ε, ανέλαβαν τα έργα των διαγωνισμών αυτών. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ξανά τους διαγωνισμούς αυτούς, ε, την πρόσκληση για υπόβλη προσφόρων για να αποφεύγουμε αυτού του είδους τις καθυστερήσεις. Για να περάσουμε στον προϋπολογισμό, όπως σας είπα, Υπάρχουν πολύ λιγότερα προβλήματα. Στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου αναφέρατε δύο σημεία. Το πρόβλημα του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΦΚΟ που πήγε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Εκτότε δημιουργήθηκαν διάφορες σύνδεσεις μεταξύ των δύο αυτών θεσμικών οργάνων. Για να σας υπενθυμίσω ήδη το 2010 υπήρξε μια απόφαση της Κομισιόν για τις αντιπροσωπείες για τη συμβάση του προσωπικού και γίνονται διαρκώς συζητήσεις μεταξύ της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης μέσω διαφορών μέσων. Στο τέλος του 2011, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει παραπάνω, η Γενική Γραμματέας της Κομισιόν, η κυρία Κατρέντε και ο κύριος Ντέβιτ Σέλβαν της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, συνυπέγραψαν ένα έγγραφο όπου δίνουν οδηγίες στις αντιπροσωπείες για τη χρήση του προσωπικού ώστε να αποφεύγεται ότι η μία από τις δύο, ο ένας από τους δύο οργανισμούς χρησιμοποιεί υπερβολικά πολύ το προσωπικό του άλλου. Θα έχουμε λοιπόν τα αποτελέσματα από τις εκθέσεις EMR του 2010 που θα μας έρθουν λίγο καιρό. Για να ολοκληρώσω αυτή τη γενική παρουσίαση, μια κοινή απόφαση μεταξύ Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και Κομισιόν ελήφθη το Μάρτιο του 2012 για το μηχανισμό συνεργασίας που αφορά τις αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια απόφαση του ΟΙΤΕΛ Προχωράνε λοιπόν τα πράγματα, αποκομίζουμε κάποια διδάγματα, θα αποκομίσουμε κάποια διδάγματα φέτο, αναμένοντα τα αποτελέσματα από τι εκθέσει των αντιπροσωπιών. Και πιστεύω θα τα δούμε αυτά τα αποτελέσματα στην έκθεση δραστηριοτήτων του 2012. Τέλο, όσον αφορά του μετρήσιμου δείκτε. Δεν κατάλαβα καλά για το αν μιλάτε για τους γνωστούς δείκτες κλειδιά που υπάρχουν στο EMR. Όπως σας είπα και προηγουμένως, από αυτό το πρώτο έτος εμπειρίας θα πρέπει να αναθεωρήσουμε μια σειρά αυτών των δικτών. Ορισμένοι πρέπει να διευκρινιστούν καλύτερα, κάποιοι άλλοι μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα, κάποιοι άλλοι θα πρέπει να επανακαθοριστούν διότι οδηγούν σε έλλειψη συνοχής. Προβλέπετε λοιπόν μια σειρά εργασιών στην Κομισιόν ώστε να είναι πιο χρήσιμοι αυτοί οι δείκτες. Το 2013 ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις που μου έθεσε ο κ. Σίγητης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Τώρα το λόγο έχουν τα μέλη. Ε, κύριε Μπέρμαν. Ευχαριστώ, Madame la Είμαι Je suis Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που έχει σταθεροποιηθεί το ποσοστό σφάλματος τα τελευταία 10 χρόνια. Αλλά όπως βλέπετε και τα μαλλιά μου σταμάτησαν να πέφτουν τα τελευταία 10 χρόνια. Σταθεροποιήθηκε η διαδικασία. Καλό θα ήταν λοιπόν να πέσει κι άλλο το ποσοστό αυτό. Με ικανοποιούν αρκετά οι απαντήσεις σας, αλλά θα μπορούσα ίσως να έρθω κάποια στιγμή να έρθω να σας δω και να συζητήσουμε όσον αφορά τις προόδους, ε, όσον αφορά τον ορισμό αυτών των δικτών, όλα αυτά τα ζητήματα πολυτεχνικής φύσης, λεπτο, σε, που αφορούν μικρές λεπτομέρειες, ώστε να μπορούσαμε να οργανώσουμε κάποια συνάντηση για να τα συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Ε, έθεσε και διάφορες ερωτήσεις η Σάσκια Μπράουν, ε, ε, διοικητικό μας εδώ και θα θέλαμε να σας ξανασυναντήσουμε αν συμφωνείτε σε μεταγενέστερο στάδιο. Πρόεδρος, παίρνω και εγώ το λόγο και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Κόρτες Λάστρα. Σημείωσα από την παρουσίαση της Κομισιόν ότι δεν είστε σε θέση να είστε βέβαιοι ότι πληρώνονται οι στρατιώτες της Μισόμ, διότι αυτό γίνεται μέσω της Αφρικανικής Ένωσης. Έχετε διενεργήσει ελέγχους. Δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να στείλετε κάποιον τις ε, ημέρες ε, ε, πληρωμής να παρατηρήσετε τι γίνεται, να ρωτήσετε διότι εκεί υπάρχει μια πηγή σημαντική διαφθοράς. Είναι ψηλέ οι αποζημιώσεις σε σχέση με το, τους μισθούς περιοχής και υπάρχει μια ε, τάση σίγουρα κάποιοι να παρακρατούν ποσά από αυτού του μισθού. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κατά πόσο γίνονται έλεγχοι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι μισθοί αυτοί καταλήγουν στου δικαιούχου του. Ο κύριο Κόρτε Λάστρα. Ναι, Πρόεδρε, μία μόνο ερώτηση θα ήθελα να διατυπώσω προς την Επιτροπή, Πρόεδρε. Ο αρμόδιος της Επιτροπής μας είπε ότι θα υπάρξει κίνηση προσωπικού στις αντιπροσωπίες ε, της Ένωσης και εξαρτάται από το πού θα υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες για αυτές τις μεταθέσεις. Αυτό ανέφερε σχολιάζοντας το. Θα ήθελα τώρα να ξέρουμε πού είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες στις ανθρωπιστικές καταστάσεις, στις ανθρωπιστικές ανάγκες, σε αναφέρεστε σε κάποιο αριθμό προγραμμάτων ή σχεδίων. Θα πρέπει να το κάνετε όμως αυτό με μεγάλη προσοχή. Εφιστώ την προσοχή της Επιτροπής σε αυτό το θέμα. Υπάρχει κίνδυνος ότι με αυτή τη μετάθεση προσωπικού θα μπορούν να υπάρχουν επιπτώσεις για κάποιες χώρες με τις οποίες έχουμε σχέση, πρέπει να έχουμε πολύ σημαντική σχέση σε σχέση με τη συνεργασία και την ανάπτυξη. Και αυτό θα μπορούσε να εκπροσωπεί ανεπαρκώς την Ένωση και να δημιουργηθούν προβλήματα στο μέλλον. Ανεξάρτητα από το πώς θα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες, ζητώ επίσης να είσαστε πολύ προσωπικοί στην κίνηση προσωπικού, να μην υπάρξουν ανισορροπίες που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν προβλήματα και να καταλήξουμε σε μεγαλύτερα ποσοστά στο μέλλον. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην Κομισιόν. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω ουσιαστικά τρεις ερωτήσεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να συναντηθούμε με τα μέλη της Επιτροπής σας για να συζητήσουμε τους δείκτες, αλλά προτείνω να περιμένουμε το δεύτερο εξάμεινο του έτους ώστε να μπορέσουμε να αναλύσουμε πρώτα σε εμά όλους τους δείκτες, να προτείνουμε βελτίωση και μετά να συζητήσουμε μαζί σας. Καλό θα ήταν λοιπόν να γίνει αυτή η συνάντηση μετά από το καλοκαίρι. Όσον αφορά του στρατιώτε, το 2012 δώσαμε εντολή για ανεξάρτητο οικονομικό έλεγχο εκ μέρου μα και ζητήσαμε ε, ελέγχου σε περισσότερο βάθο από την Αφρικανική Οργάνωση. Αντιλαμβάνομαι το αίτημά σα. Πρέπει οπωσδήποτε να προσφέρουμε αυτή τη διασφάλιση, αλλά χρειάστηκε να περιμένουμε να περάσει κάποιο χρόνο λειτουργία και τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή για αυτόν τον οικονομικό έλεγχο. Όσον αφορά την ανακατανομή του προσωπικού, επιμένω μιλάμε για προσωπικό που εξαρτάται από την DEVCO, όσο αφορά δηλαδή την ανάπτυξη, όχι το σύνολο του προσωπικού. Σαφώς λοιπόν σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, για παράδειγμα σε αναδυόμενες χώρες στην Ασία, για παράδειγμα στην Ινδία όπου υπήρξε τεράστια συνεργασία, δεν υπάρχει πια λόγος για αυτή τη συνεργασία. Εκεί λοιπόν σε θέματα ανάπτυξης, θα μειώσουμε την αρρωγή προς την Ινδία, το ίδιο και στην Κίνα, όπου είχαμε πολύ κόσμο και αυτό το ανθρώπινο δυναμικό που θα φύγει από αυτές τις αντιπροσωπείες θα ανακατανεμηθεί σε αντιπροσωπείες που το χρειάζονται περισσότερο. Συνήθως μιλάμε για την υποσαχάρια Αφρική και τις γειτονικές περιοχές όπου βλέπουμε να εμπλουτίζεται το πρόγραμμα η ανακατανομή λοιπόν σχετίζεται με τον επαναπρογραμματισμό υπό την ε, αιγίδα της ΔΕΒΚΟ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπέρμαν. Όχι, όχι, εγώ είπα όσα είχα να πω. Σας ξαναδίνω το λόγο με μεγάλη ευχαρίστηση. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι η προθεσμία είναι 24 24η Ιανουαρίου 5 το απόγευμα για την κατάθεση των τροπολογιών και η ψηφοφορία θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου. Θα περάσουμε τώρα στο σημείο 10 τον κανονισμό για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Σώματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ θα μας παρουσιάσει τις εμπειρίες που έχει από τα πιλωτικά προγράμματα για την εθελοντική προσφορά. Τα εθελοντικά προγράμματα <clears throat> λειτουργούν από το 2011 και μετά και οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να καταλήξει σε πολύτιμα θα έλεγα συμπεράσματα σχετικά με την πιθανότητα δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών όπως μας γνωστοποιήθηκε στις αρχές του χρόνου. Να πω επίσης ότι η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ θα μας παρουσιάσει μέσω του κυρίου Χένκ τις εμπειρίες της. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα στην συνεδρίασή σας. Είμαι το σημείο επαφής για τους εθελοντές στο εσωτερικό της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ. Θα σας παρουσιάσω κάποια από τα μαθήματα στα οποία καταλήξαμε μέσω της πιλωτικής φάσης. Ξέρετε ότι συνήθως εμείς κάνουμε τρία χρόνια προπαρασκευαστικής βάσης πριν τεθεί σε λειτουργία η νομική βάση θα έλεγα και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα μαθήματα λοιπόν που πήραμε από τη διαδικασία αυτή και το πώς τροφοδότησαν οι εμπειρίες αυτές τον κανονισμό που είναι υποσυζήτηση. Θα υπάρξουν πολλές παραπομπές στις διαφάνειες τις οποίες θα δείτε σχετικά με το αρχικό κείμενο του κανονισμού. Βλέπετε εδώ μια περίληψη του τριετούς προγράμματος, τα βασικά χαρακτηριστικά στα οποία εμείναμε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι το 2011 συγκεντρώσαμε την προσοχή μας σε νέους εθελοντές, άπειρους, το άπειρο κομμάτι των ενδιαφερομένων εθελοντών, μείωση κινδύνου, πρόληψη και ε, ανάκαμψη μετά το τέλος της κρίσης. Αυτά είναι τα πρώτα πιλωτικά προγράμματα του 11. Το 12 διευρύναμε την εμβέλεια των προγραμμάτων αυτών στην ε, ικανότητα ίδιας ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο και στην αύξηση της αντοχής των πληθυσμών. Το 2013 προβλέπουμε να συμμετέχουν και κάποιες χώρες και εθελοντές από τρίτες χώρες. Και έχουμε όχι μόνο με μονομένους εθελοντές, αλλά και ομάδες εθελοντών. Σήμερα ή αύριο, ανάλογα πόσο γρήγορα θα πάει η διοίκηση, θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός για το 2013 και εδώ έχουμε τους λεγόμενους εμπειρογνώμονες εθελοντές, όχι μόνο τους νέους που ελέγξαμε το 11 και το 12, αλλά εθελοντές με συγκεκριμένη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη την οποία θα απαιτήσουμε. Και ο δεύτερος στόχος μας για τα πιλωτικά του 13 θα είναι οι δυνατότητες ε, ε, βοήθειας τοπικής ανάπτυξης. Ξέρετε ότι έχουν γίνει πολλές συζητήσεις με ανθρωπιστικές οργανώσεις και αυτού του προγράμματος βασικό τμήμα θα πρέπει να είναι η ίδια δυνατότητα ανάπτυξης. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι έχουμε άνω των 200 εθελοντών που έχουν πάει σε διάφορες χώρες πάνω από 30 χώρες εκπροσωπούνται στα πλαίσια αυτού του ε, προγράμματος, 40 οργανώσεις που είναι εταίροι ή συμμετέχοντες και εκπροσωπούν 19 χώρες μέλη. Όλα αυτά τα αρχικά τα σήματα που βλέπετε είναι οι υπεύθυνοι ε, για τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται σε αυτή τη φάση. Εδώ είναι ένας χάρτης ε, των χωρών στις οποίες έχει αναπτυχθεί η βοήθειά μας τα τελευταία χρόνια. Το νέο κύμα των εθελοντών τώρα θα πρέπει να ε, μπει και αυτό στον πίνακα, αλλά εδώ βλέπετε βασικά τις χώρες στις οποίες έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν οι εθελοντές μας. Καλύπτουμε όλες τις υπήρους και ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί των χωρών μετά το 2013. Αυτό το οποίο θελήσαμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης είναι να οργανώσουμε πολλές συναντήσεις με τους συντονιστές ε, των ε, συγκεκριμένων προγραμμάτων συζητήσαμε μαζί τους τα μαθήματα στα οποία κατέληξαν από τις εμπειρίες τους και εμείς προσπαθήσαμε από τα προγράμματα αυτά να δούμε εξ αρχής τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Επισκεφθήκαμε και τα περισσότερα από τα προγράμματα αυτά, έτσι λοιπόν είδαμε τους εθελοντές πριν να φύγουν για τις αποστολές τους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περίοδου και είχε και επαφή και η Επίτροπος Γεωργίευα για να δούμε τι, να δει τι συμβαίνει σε σχέση με την πείρα που συλλέγουν αυτά τα άτομα. Και φυσικά όλες αυτές οι οργανώσεις δεν σταμάτησαν στο να μας λένε ποιες είναι οι απόψεις τους για αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε πολλές τέτοιες παρεμβάσεις που έγιναν από τα μαθήματα τα οποία έχουν συναχθεί από αυτή την πρωτοβουλία. Αυτά οδηγούν σε αυτό το οποίο θα παρουσιάσω τώρα. Και όπως είπα πάντα θα προσπαθώ άμεσα να συνδέω τα μαθήματα τα οποία έχουμε συναγάγει με το πώς εφαρμόστηκαν αυτά υπό τον κανονισμό. Δεν είναι το καλύτερο σε σχέση με το πράσινο. Βλέπετε αριστερά και δεξιά. Αριστερά ποια τα μαθήματα και τι κάνουμε με αυτά τα οποία συνήθισαν ως συμπεράσματα. Και είναι τα άρθρα ή τα εδάφια στον κανονισμό οι αριθμοί. Πρώτο μάθημα. Υπάρχει μεγάλη υψηλή ζήτηση νέων εθελοντών να προσχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Αυτό που ακούσαμε πολύ συχνά είναι ότι οι εθελοντέ και αυτό το πρόγραμμα φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένο για του νέου που θέλουν να εμπλακούν στον τομέα αυτό και που όμω ακόμα δεν έχουν την πείρα, την επαγγελματική πείρα και την επαγγελματική πείρα επιτόπου ώστε να μπορούν να εργαστούν επιτόπου σε τέτοιο πρόγραμμα ή σχέδιο και να επιλεγούν από τι ανθρωπιστικέ οργανώσει. Ανθρωπιστικές οργανώσεις επιλέγουν πεπειραμένα άτομα που έχουν ήδη προηγούμενη πείρα. Και εδώ σε σχέση με αυτούς τους ε, εθελοντές υπάρχει η θετική προσθετή αξία. Γι' αυτό στο δεξί χέρι βλέπετε ότι στον κανονισμό δεν έχουμε ένα ελάχιστο ή μέγιστο για την ηλικία. Θέλουμε να είμαστε ελαστικοί και να είμαστε ανοιχτοί για τους νέους εθελοντές που θέλουν να εισαχθούν στον τομέα, να, μπορέσουν να μπουν σε αυτόν τον τομέα και σε σχέση με τις 6.400 τέτοιες δράσεις που προβλέπονται για την επταετή αυτή η περίοδο, έχουμε ένα υψηλό ποσοστό υψηλής ε, ε, μακροπρόθεσμης ε, δραστηριότητας και ένα χαμηλότερο ποσοστό βραχυπρόθεσμης δράσης που θα είναι μάλλον πιο ενδιαφέρουσα για τους πεπειραμένους εργαζόμενους που έχουν ήδη συλλέξει πείρα και έχουν και τη δυνατότητα να πάνε στην Αλαδαπή. Γιατί έχουν επιλεγεί αυτοί οι νέοι εθελοντές που είναι ενδιαφέρον αυτό το εγχείρημα. Ακούσαμε και ιδιαίτερα από τις οργανώσεις ε, του τομέα ότι αυτό που επίσης χρειάζονται είναι οι δεξιότητες, οι πεπειραμένοι εθελοντές. Δεν κλείνουμε την πόρτα σε αυτούς, όμως προβλέπουμε επιμερισμό των, του έργου σε σχέση με τα εθελοντικά αυτά προγράμματα εθελοντών, επιμερισμό έργου. Αυτό το οποίο ε, έχει αρκετά συχνά αναφερθεί είναι ότι δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στην δράση επιτόπου, αλλά και για την ε, ε, επιμελητιακή υποστήριξη. Αυτά μπορούν να τα κάνουν πολλές φορές οι εθελοντές χωρίς να πάνε σε μια τρίτη χώρα. Ε, στο διαδίκτυο, online, online volunteering, δηλαδή διαδικτυακή εθελοντική δράση που είναι ένα, μια άλλη συνιστόσα αυτής της προσπάθειας. Αν δούμε την επιλογή και την στελέχωση, την επιλογή για τα στελέχη αυτά, εκπληκτικός αριθμός ε, έχει παρουσιαστεί. 100 υποψήφοι για μία τέτοια τοποθέτηση ε, στην Ισπανία με τις ισπανικές οργανώσεις που προσέλαβαν τις τελευταίες εβδομάδες ένα πολύ μεγάλο αριθμό που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως έργο και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιο μεγάλο αριθμό ατόμων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και φυσικά αυτό το οποίο εντάξαμε, εντάξαμε στον κανονισμό είναι ότι δεν είναι σίγουρα μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την το χτένισμα των ε, ε, υποψηφιωτήτων, οι οργανώσεις θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της δράσης, να μπορούν να επιλέγουν τα άτομα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τα οποία τους ενδιαφέρουν. Επίσης ενδιαφερόμαστε για, ένα ε, μια προσέγγιση από πλευράς κανονισμού για ένα συγκεκριμένο μητρό. Όταν βλέπει κανεί τι γίνεται με τα μητρώα των κρατών μελών, για παράδειγμα, όπου μπορούν να αυτοκαταχωρηθούν τα άτομα και να περιμένουν να δουν αν θα ζητηθεί να ε, δραστηριοποιηθούν στο μέλλον. Αυτό δημιουργεί πολλέ προσδοκίε και πολλέ φορέ αν δεν υλοποιηθούν αυτέ οι ε, προσδοκίε, ε, απογοήτευση. Αυτό που σκεφτήκαμε εμεί είναι με την καταχώρηση αυτή μόνο άτομα τα οποία έχουν επιτυχώς επιλεγεί από έναν αποστέλλοντα οργανισμό και έχουν καταρτιστεί και έχουν αξιολογηθεί ως κατάλληλα άτομα για τέτοια αποστολή, μόνο αυτά θα καταχωρούνται σε τέτοιου είδους μητρώα. Αυτό σημαίνει σημαντική διαδικασία ε, χτενίσματος όσον αφορά για παράδειγμα ένα κοσκίνισμα τέτοιων υποψηφιωτήτων για να μπορούν να είναι τα κατάλληλα άτομα που θα χρησιμοποιηθούν και θα επιλεγούν. Είμαστε ιδιαίτερα, έχουμε ιδιαίτερα υπόψη ότι πρέπει να υπάρχει ε, δίκαιος χαρακτήρας όσον αφορά την επιλογή Κάποιοι εθελοντέ ή κάποιοι που δεν επελέγησαν είπαν ότι καμιά φορά είναι θολή η διαδικασία, αδιαφανή. Αν αφήνουμε έναν οργανισμό να επιλέγει, για παράδειγμα, ποιοι θα είναι οι εθελοντέ αυτέ, όπω γίνεται για τέτοιου είδου εθελοντικά προγράμματα, πρέπει να ξέρουμε πώ επιλέγονται σε σχέση με τι προδιαγραφέ που θεσπίζονται. Να μην έχουν του δικού του ή τα δικά του στελέχη ε, με τα οποία έχουν επαφέ τέτοιου είδου οργανώσει, αλλά να είναι ανοιχτό ένα τέτοιο πρόγραμμα σε όλου που ενδιαφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα είναι ένα στοιχείο των προδιαγραφών που θα θεσπίσουμε ώστε να υπάρχει αυτή η διαφάνεια. Επίση είδαμε στα σχέδια για το 2011 μεγάλο αριθμό αποτυχόντων εθελοντών. Εθελοντών που δεν ολοκλήρωσαν δηλαδή αυτό το πρόγραμμα μέχρι τέλους. Μπορείτε να το δείτε αυτό και σαν αρνητικό αλλά και σαν θετικό στοιχείο. Γιατί τι συνέβη για αυτούς που έφυγαν, αποχώρησαν, βρήκαν μια θέση επιτόπου αμέσως. Είμαστε θύματα της ίδιας επιτυχίας μας μέσα από αυτό για παράδειγμα. Αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιούνται τα προγράμματα θα αποτελεί τη βέλτιστη χρήση των κονδυλίων. Δεν θα καταρτίζουμε εμείς με αυτά τα κονδύλια και μετά από λίγο τα καταρτισμένα αυτά εξειδικευμένα άτομα θα αποχωρούν. Πρέπει η επένδυση στα άτομα αυτά να διασφαλίζει ότι τα άτομα αυτά θα παραμένουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και θα υπάρχει μια προοπτική μετέπειτα για τέτοιου είδους σταδιοδρομία. Επόμενο. Ένα από τα σημεία που όλοι οι εμπλεκόμενοι ανέφεραν και είναι πολύ σημαντικό είναι φυσικά το εμπόριο. Και είδαμε σε σχέση με την κατάρτιση, την κατάρτιση διορθώνω, το τι πρέπει να γίνει και συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να υπάρχει σε βάθος προετοιμασία για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τέτοιες δράσεις. Οι ανθρωπιστικές δράσεις δεν είναι ε, κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά και για τις πτυχές της ασφάλειας. Να ξέρει κανείς πού πηγαίνει και σε ποιο μέρος θα πάει και να ξέρει πώς πρέπει να αντιδράσει. Κατάρτιση, εκπαίδευση ε, θα πρέπει να, να την χάνει ιδιαίτερης προσοχής οι περισσότεροι χρησιμοποιούν ε, συνδυασμένη προσέγγιση, διαδικτυακή εκπαίδευση και κατάρτιση και επιτόπου εκπαίδευση και κατάρτιση όταν ε, συλλέγονται και βρίσκονται επιτόπου οι επιλεγέντες ε, εθελοντές. Πρέπει εδώ να δούμε πώς όλα αυτά θα μεταφράζονται στο ότι θα έχουμε προβλέψει και θα έχει γίνει η πρόβλεψη για υψηλό αριθμό για την κατάρτιση. 5-6 για παράδειγμα ευρώ για τέτοιου είδους ε, κατάρτιση εκπαίδευση είναι σχετικά υψηλό ποσό για τέτοιες δράσεις. Επίσης, οι ανθρωπιστικέ οργανώσεις ήθελαν ιδιαίτερα εμείς να συμπεριλαμβάνουμε για αυτές μια δυνατότητα αξιολόγηση των εθελοντών που αποστέλλονται. Κάτι το οποίο συμπεριλάβαμε λοιπόν στον κανονισμό είναι μια τοποθέτηση μαθητείας εντός εισαγωγικών. Έτσι, η εξοικείωση από αυτά που ακούσαμε από τις οργανώσεις, αν θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούν να αποσταλούν τέτοιου είδους νέοι εθελοντές, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα της κατάρτισης εκπαίδευσης αξιολόγησης αυτών των εθελοντών εδώ στην Ευρώπη, προτού αποσταλούν στο πεδίο δράσης επιτόπου. Γι' αυτό έχει, έχουμε καταλήξει σε αυτό τον υψηλό αριθμό 2.300 ατόμων προς μαθητεία και κατάρτιση που πρώτα στο επιτελείο μας θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να καταρτιστούν προτού αποσταλούν επιτόπου προς δράση ως εθελοντές. Οι ίδιοι οι εθελοντές ενδιαφερόντουσαν ιδιαίτερα για τη διαπίστευση, ώστε στο ε, βιογραφικό τους να μπορεί να ξεχωρίζει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε προβλέψει σε κάποια εδάφια και είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα αποτελεί τμήμα των προδιαγραφών και απαιτήσεων θα απαιτήσουμε, θα ζητηθεί από τέτοιες οργανώσεις να προβλέπονται τέτοιες δυνατότητες, ώστε να παίρνουν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις οι εθελοντές, ώστε να έχουν ένα κάτι το οποίο θα έχουν στα χέρια τους ως κεκτημένο για, για αυτή τη δραστηριότητα στο βιογραφικό τους μετέπειτα. Και καταλήγω τώρα σε ένα σημείο το οποίο βλέπετε εδώ με κόκκινο, και που είναι πιο ανάγλυφο και πιο ευδιάκριτο. Σίγουρα θα ακούσατε και θα παρατηρήσατε συζητώντας τα θέματα αυτά για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις ένα σημείο όπου δεν συμφωνούμε αναγκαία με, αυτή την, ε, με αυτές τις οργανώσεις είναι ότι θέλουν αυτές οι ίδιες να διοργανώνουν αυτή την κατάρτιση και εκπαίδευση οι ίδιες και όχι εμείς η Επιτροπή που θα παρέχει η κατάρτιση σε συγκεκριμένα θέματα. Γιατί λοιπόν εμείς ε, προβληματιστήκαμε και σκεφτήκαμε να το προσεγγίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το οποίο είδαμε οπωσδήποτε είναι θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε θελοντή που θα περνάει από αυτή τη διαδικασία θα, έχει, θα την χάνει τη ίδια κατάρτιση και εκπαίδευση και θα καταλήγει στο ίδιο επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Αν δείτε τι διαφορετικέ οργανώσει ε, με τι οποίε συνεργαστήκαμε, κάποιε έχουν ισχυρέ επιδόσει, άλλε όχι τόσο ισχυρά δυνατά προγράμματα. Για να υπάρχει ισότιμη λοιπόν τέτοια δραστηριότητα για όλους τους εθελοντές πρέπει να μπορούν να ακολουθήσουν τα ίδια μαθήματα και την ίδια σχετική κατάρτιση. Και ένα άλλο θέμα το οποίο ε, προσεγγίζουμε είναι ότι υπάρχει αξία στο να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή κατάρτιση όπου θα συνέρχονται εθελοντές από διαφορετικά προγράμματα. Γιατί διαφορετικά θα έχουμε προγράμματα του Ερυθρού Σταυρού, του Save the Children, ώστε ε, να σώσουμε τα παιδιά προγράμματα και θα υπάρχει διαφορετική ας το προσέγγιση. Είδαμε ότι η αρχική περίοδος κατάρτισης είναι η στιγμή εκείνη που μπορούν να συνέρχονται από διαφορετικά προγράμματα οι εθελοντές που θα θεωρούν ότι είναι μέρος και τμήμα κοινού προγράμματος και θα δημιουργείται το πνεύμα εκείνο του να ανήκει κανείς σε μία μονάδα ή σε ένα σώμα, esprit de corps. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτοματισμός θα έλεγα σε σχέση με τις οργανώσεις αυτές για τη διαμόρφωση της κατάρτισης. Όμως θα υπάρχει ένας τέτοιος ε, ανοιχτός χαρακτήρας υποβολής προσφορών ε, ή ε, διαμόρφωσης των προγραμμάτων κατάρτισης, π.χ. για τον Ερυθρό Σταυρό, ώστε να υπάρχει πριν από την δραστηριοποίηση των εθελοντών εθελοντών δυνατότητα να παρέχεται επιπρόσθετη κατάρτιση πέρα από αυτή που θα παρέχουμε εμείς για, για εκείνα τα πεδία που θεωρούν ενδεδειγμένα οι οργανώσεις αυτές όπως π.χ. ο Ερυθρός Σταυρός. Και εδώ το θέμα της αναφοράς των οργανώσεων υποδοχής και των σωμάτων των οργανισμών που αποστέλουν τέτοιους εθελοντές πρέπει να διασφαλίσετε το υψηλό επίπεδο πείρας και δεξιοτήτων ώστε να γνωρίζουμε ποιος είναι εκείνος ο οποίος αποστέλλεται. Οι Ευρωπαίοι εθελοντές να μπορούν να έχουν τη σωστή αντιμετώπιση όσα συσχετίζονται με την ασφάλεια, το καθήκον περίθαλψης, ε, την ε, ε, παρακολούθηση και την ε, ε, αρρωγή, πληρωμές, μισθή, άδειες. Όλα αυτά θα αποτελούν τμήματα των προδιαγραφών των διατάξεων που θα εκπονηθούν. Ακόμα και αν όλα αυτά ακόμα δεν βρίσκονται εξειδικευμένα στο επίπεδο κανονισμού, διότι είναι πολύ εξειδικευμένα θέματα, θα εκπονήσουμε τέτοιου είδους ε, ε, διατάξεις ώστε να αποτελούν μέρος των συμβάσεων που θα συνάπτουν οι εθελοντές ατομικά με τον αποστέλλοντα οργανισμό ή οργάνωση. Και ένα άλλο σημείο που στη δεξιά πλευρά θα δείτε πάλι με κόκκινο είναι η ελίπουσα, το ε, απουσιάζον νομικό καθεστώς για τα μέλη, για τα κράτη-μέλη, όπου διαφορετικά κράτη έχουν διαφορετικούς κανόνες και κανονισμούς όταν έχουμε την εμπλοκή διεθνών εθελοντών. Κάποιες χώρες δεν έχουν καν κανόνες ε, για αυτούς. Ε, και σε σχέση λοιπόν με το νομικό καθεστώς αυτών των εθελοντών ε, υπάρχουν ίσως ενδεχόμενα κενά. Αυτό είναι κάτι που σε σχέση με τον κανονισμό δεν μπορέσαμε να επανορθώσουμε και να καλύψουμε αυτό το κενό, αυτή την έλλειψη. Διότι από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έπρεπε να γίνει η προσπάθεια να εξευρεθεί ένα κοινό καθεστώς για αυτούς τους διεθνείς εθελοντές που θα μετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το ε, αξιολογούσε ιδιαίτερα ο τομέας αυτός. Και σε σχέση σε, και με τις απολαβές ε, έπρεπε κάποια στοιχεία να επινοήσουμε πώς θα πληρώνονται τέτοιου είδους ε, ε, θα πληρώνονται μισθοί, ώστε να δούμε πώς θα φορολογούνται. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, αλλά είναι σημαντικό για τους εθελοντές να έχουν ένα αναγνωρισμένο νομικό καθεστώς. Δυστυχώς αυτό υπεκφεύγει του εύρους του, του πλαισίου του κανονισμού, πρέπει όμως να το έχουμε υπόψη ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί όπως πρέπει στο μέλλον. Ένα ενδιαφέρον σημείο που επανέρχεται σε όλα τα έργα είναι η κότα και το αυγό. Δηλαδή πρώτα να επιλογούν οι εθελοντές ώστε οι οργανισμοί φιλοξενίας υποδοχής να βρουν θέσεις κατάλληλες για τους εθελοντές ή πρέπει να υπάρχουν πρώτα οι θέσεις να έχουν προκηρυχθεί και μετά να ξέρουμε για ποια θέση προσλαμβάνουμε ποιον. Διότι πολύ συχνά οι εθελοντές δεν θέλουν να κάνουν αίτηση ε, στα τυφλά θέλουν να ξέρουν γιατί αιτούνται, αλλά και οι οργανισμοί από την άλλη δεν θέλουν απαραίτητα να ανοίξουν μια θέση χωρίς να γνωρίζουν ποιος εθελοντής θα ε, καταλάβει αυτή τη θέση. Αυτό το απαντήσαμε στον κανονισμό λέγοντας ότι η αξιολόγηση αναγκών είναι αυτή που πρέπει να λαμβάνει η χώρα πρώτα, δηλαδή Πρώτον, οι οργανισμοί υποδοχής πρέπει να γνωρίζουν τις ανάγκες της κοινότητας του οργανισμού υποδοχής και μόνο τότε θα ε, ανακοινώνουν ε, καινέ θέσεις. Αυτό είναι κάτι λοιπόν που επανεξετάσαμε και σίγουρα είναι κάτι που αποτελεί αρχή στην ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει πρώτα να έχουν καθοριστεί οι ανάγκες ε, πριν παρασχεθεί η αρρωγή. Θέλω να τονίσω ότι όπως είδατε στο πιλωτικό έργο δεν έχουμε επιλέξει ακόμα έργο αντιμετώπισης καταστροφών. Όλα τα έργα μέχρι στιγμής ε, είχαν να κάνουν με μείωση κινδύνων, καταστροφής, ε, αποκατάσταση μετά από κρίση, ε, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, αλλά όχι πραγματική απόκριση σε περίπτωση καταστροφής. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι φυσιολογικό, διότι μέχρι στιγμής εστιαστήκαμε σε νέους και άπειρους εθελοντές. Τώρα, στα έργα του 2013, Αυτά απευθύνονται κυρίω σε εξειδικευμένου εθελοντέ με τεχνική εμπειρία και θα δούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε Φέτο να έχουμε κάποιο έργο για αυτό το συγκεκριμένο πεδίο. Δεν το έχουμε αποκλείσει στον κανονισμό, Μα επιτρέπει να περιλαμβάνουμε την απόκριση σε περίπτωση καταστροφή, παρότι ορισμένοι λένε ότι πρέπει να στείλουμε οπωσδήποτε ανθρώπου που ξέρουμε ότι μπορούν να παρέχουν αποτελέσματα για μα. Αυτοί είναι οι έμπειροι εθελοντέ. Βλέπω ότι περνάει ο χρόνο. Δεν θα μπω λοιπόν σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα να τονίσω ένα σημείο. Για ποιο λόγο αναφέρθηκε αυτό στον κανονισμό η ανάπτυξη σε γραφεία της ΕΚΟ. Έχουμε συμπεριλάβει αυτή τη δυνατότητα, δεν έχει εφαρμοστεί, διότι δεν γίνεται να ε, στέλνουν οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί εθελοντές σε γραφεία της ΕΚΟ και είναι δύσκολη χρηματοδότηση αυτού διότι φυσικά οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί πρέπει να παρέχουν συγχρηματοδότηση για την αποστολή εθελοντών σε γραφείο της ΕΚΟ και η παροχή τέτοια συγχρηματοδότησης δημιουργεί ένα περίεργο καθεστώ. Αυτό που συμπεριλάβαμε λοιπόν στον κανονισμό είναι το εξή ότι στέλνει η Κομισιόν ανθρώπινο δυναμικό σε γραφεία τη Κομισιόν. Εάν υπάρχει λοιπόν μικρό αριθμό εθελοντών που θα σταλεί σε γραφεία της Επιτροπής. Αυτό θα γίνει από την ΕΚΟ και όχι από τους μη κυβερνητικού οργανισμούς. Το είπαμε λοιπόν ευθέω ώστε να μην περιπλέκουμε την κατάσταση. Μια σαφή έκκληση από όλου του οργανισμού ήταν ότι η ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού που έχει ήδη αναφερθεί, θα δείτε στο άρθρο 15, ανοίγει ένα τεράστιο εύρο δυνατοτήτων για την ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού. Δηλαδή, δεν θα επενδύουμε μόνο στου εθελοντές από την Ευρώπη αλλά και σε τοπικό ανθρώπινο δυναμικό. Και θα κλείσω με κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, την οποία φυσικά προσπαθούμε να καθιερώσουμε με αυτό το πρόγραμμα. Είναι βέβαιο και έχει διαπιστωθεί στα πιλωτικά έργα, εμπλέκονται πολλοί οργανισμοί, πάνω από 40. Μιλάμε τώρα για συνεργασίες οι οποίες διαμορφώνονται μέσω των πιλωτικών έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν προϋπήρχαν. Για ένα παράδειγμα, το Save the Children έκανε ένα έργο μαζί με πανεπιστήμια, με την Bioforest που είναι ένα γαλλικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτό, όπως μας είπαν οι διάφοροι αυτοί οργανισμοί, κοστίζει χρόνο και επενδύσεις και είναι λίγο δυνηρό, διότι οι συνέργειες αυτές δεν είναι απαραίτητα αποτελεσματικές. Από την άλλη όμως, Πρόκειται για συνεργασίες που αναδεικνύουν τις καλύτερες πρακτικές του τομέα, διότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί έχουν αναπτύξει βέλτιστες πρακτικές του τομέα τους και μόνο μέσω αυτών των συνεργασιών μπορούμε να ε, αναδείξουμε όλες τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτή είναι λοιπόν μια προσθέμενη αξία κατ' εμάς στην πιλωτική φάση και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει και προσθέμενη αξία για το τελικό πρόγραμμα. Γι' αυτό την έχουμε συμπεριλαβεί ως γενική αρχή αυτή τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ συμμετεχόντων οργανισμών στο πρόγραμμα. Τέλος, όσον αφορά την ευρωπαϊκή ε, προσθέμενη αξία, αυτό το ομαδικό πνεύμα και η οικοδόμηση ταυτότητας στο πρόγραμμα. Αυτό που ακούω συχνά από εθελοντές στα πιλωτικά έργα μου λένε τι είναι αυτό το πρόγραμμα, γιατί ανήκω εγώ σε αυτό, γιατί δεν βλέπω εθελοντές από άλλα προγράμματα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι σχετικά δύσκολο να το αντιληφθεί κανεί στι πιλωτικέ φάσει, διότι ακόμα οι διάφορε δυνατότητε βρίσκονται υποδοκιμή. Αλλά στο τελικό πρόγραμμα αυτό που σίγουρα θέλουμε είναι να μην είναι ένα πρόγραμμα που θα στέλνουμε εθελοντές εκεί όπου έχουμε πολλούς. Θέλουμε να είναι ένα πρόγραμμα που θα συναντώνται διάφοροι Ευρωπαίοι εθελοντές σε διάφορα κομμάτια του προγράμματος κατά την κατάρτιση ή κατά την ανάπτυξη και θα φροντίσουμε να μεριμνήσουμε για τη δικτύωση αυτών των εθελοντών που συμμετέχουν. Κατά τη διάρκεια δηλαδή του προγράμματος αλλά και μετά το πρόγραμμα θα υπάρχει αυτή η επαφή μεταξύ εθελοντών με τους, επαφή με τους τρέχοντες εθελοντές που θα τους ε, παρέχουν πληροφορίες από την εμπειρία τους και έτσι δημιουργείται, διαμορφώνεται μια ταυτότητα των Ευρωπαίων εθελοντών που θα προσθέσει αξία σίγουρα σε αυτούς τους εθελοντές. Ως γενικό, κάποια γενικά συμπεράσματα, φυσικά αυτά τα πιλωτικά έργα μας προσφέρουν διδάγματα τα πιλωτικά έργα φυσικά διαρκούν ελάχιστο χρόνο για τη σύσταση των προγραμμάτων και όπως είπαν όλοι υπήρξαν χρονικοί περιορισμοί οι οποίοι υποβάθμισαν την ποιότητα των προγραμμάτων. Γι' αυτό το λόγο στο τελικό πρόγραμμα θα φροντίσουμε να υπάρξουν μακρύτερες, μεγαλύτερες, πιο μακροχρόνιες συνεργασίες ώστε να μην υψέρχεται αυτός ο παράγοντας χρονικού περιορισμού και να μην παίζει τόσο σημαντικό ρόλο επιλέξαμε μία προσέγγιση, όπως είπαμε, κινητοποίησης. Ε, ε, δεν συμπεριλάβαμε όλες τις λεπτομέρειες των προτύπων μέσα στον κανονισμό, γιατί έχουμε ακόμη να μάθουμε πολλά από τα πιλωτικά έργα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Θα, οι λεπτομέρειες θα ρυθμιστούν με κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις, ώστε να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε στα πρότυπα και στο πρόγραμμα τα διδάγματα από τι εμπειρίε μα. Και αυτό θα μα επιτρέψει να έχουμε και περισσότερο χρόνο, διότι ο κανονισμό φυσικά πρέπει να κυκλοφορήσει τώρα, αλλά τα πρότυπα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχουμε χρόνο να τα ε, δημιουργήσουμε, να τα κανονίσουμε ε, σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού υιοθετηθεί ο κανονισμό. Στην τελευταία διαφανή θα να σα δείξω αυτό που βλέπετε στην οθόνη. Όπω είδαμε, μερικέ φορέ ε, τα νούμερα δεν είναι σωστά. Τα νούμερα που κυκλοφορούν όσον αφορά τα προγράμματα δεν είναι σωστά. Εδώ έχετε τα νούμερα των δικαιούχων στα δεξιά και ένα από τα λανθασμένα νούμερα ήταν 10.000 άτομα έχουν αναπτυχθεί. Ουσιαστικά το σωστό είναι 6.400 άτομα έχουν αναπτυχθεί και 3.200 άτομα σε μαθητεία. 9.000 δηλαδή 600 όπως εμφανίζεται στον κανονισμό. Όπως βλέπετε δηλαδή ο τελικός αριθμός είναι 6.400 και όπως βλέπετε, βλέπετε εδώ και τα κόστη και τα ποσοστά χρηματοδότησης, συγχρηματοδότησης σε αυτή τη διαφάνεια. Εδώ θα ήθελα να κλείσω και σας ευχαριστώ και πάλι που μου δώσετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτά τα διδάγματα που αποκομίσαμε σήμερα. Είναι άλλοι δύο συνάδελφοί μου εδώ και φυσικά ε, είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε οποιασδήποτε ερωτήσεις σε σχέση με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω κύριο Στίφλερ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας η οποία ήταν ιδιαίτερα πλήρης και χρήσιμη και για τη δική μου έκθεση. Είχα κάποιες ερωτήσεις τις οποίες απαντήσατε όμως πριν τις θέσω. Πριν λίγο καιρό είχα συναντήσει τους 21 εθελοντές του πιλωτικού προγράμματος που οργανώθηκε από τον Γαλλικό Ερυθρό Σταυρό μετά το πέρας της αποστολής. Είχαμε επικοδομητικές ανταλλαγές απόψεων, απέκτησαν πραγματικά ικανότητες ανεκτήμητες, βοηθώντας τους πληθυσμούς που τους είχαν ανάγκη. Οι περισσότεροι των νέων που πήραν μέρος στο πιλωτικό πρόγραμμα έχουν μια γενικού τύπου εκπαίδευση και εμπειρία και ο εθελοντισμός τους επιτρέπει να μπουν στον κόσμο της εθελοντικής απασχόλησης και με επαγγελματική αν θέλετε σκοπιμότητα. Εφόσον βέβαια προσφέρουν μια επιπλέον προστιθέμενη αξία στην κοινή προσπάθεια. Ήταν σημαντικό επίσης να επιλέξουμε εμπειρογνώμονες και με τεχνικές γνώσεις και συνταξιούχους και εδώ επιμένω ιδιαίτερα Νομίζω όμως ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε στη χρησιμότητά τους. Υπήρξαν πολλαπλά προφίλ τα οποία έγιναν αντικείμενο της επιλογής. Θα πρέπει η τοποθέτηση των εθελοντών να γίνει σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες και ανάλογα με τις περιφέρειες στις οποίες θα αναλυφθούν δράσεις. Οι εθελοντές αυτοί θα πρέπει να επιλαγούν επί τη βάση των αρμοδιοτήτων τους και σε τομείς στους οποίους υπάρχουν ελλείψεις στις χώρες υποδοχές. Η επιλογή και η οργάνωση θα πρέπει να σεβαστεί και τις ικανότητες των νέων και των ηλικιωμένων και των συνταξιούχων εθελοντών και κυρίως τις γνώσεις τους. Είπατε ότι οι αποστολές οργανώνονται στα πλαίσια συγκεκριμένων πιλωτικών προγραμμάτων. Θα ήθελα να μας δώσετε κάπως περισσότερες λεπτομέρειες εδώ. Τι ακριβώς είναι αυτό στο οποίο αναφέρεστε. Στον κανονισμό λέγεται ότι η Επιτροπή διαμορφώνει ένα πρόγραμμα κατάρτισης των εθελοντών στα πλαίσια των ε, μονάδων που οργανώνουν τις αποστολές. Πώς ακριβώς προβλέπετε εσείς λοιπόν να γίνει η κατάρτιση των εθελοντών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις ΜΚΟ. Νομίζω ότι η κατάρτιση θα πρέπει να βασίζεται στους ευρωπαϊκούς και εθνικούς ισχύοντες κανόνες και σε συνεργασία με ειδικευμένα θεσμικά όργανα και με οργανώσεις ανθρωπιστικές όπως αυτές που συνάντησα την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν κάποιες από αυτές τις οργανώσεις προχωρήσει αρκετά. Είμαι ικανοποιημένη που σας άκουσα να λέτε ότι οι εθελοντές συγκεντρώνουν την προσοχή τους στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, την μείωση των κινδύνων και την ανοικοδόμηση των χωρών μετά το τέλος των καταστροφών. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία αυτό που είπατε και αυτό το σώμα των εθελοντών θα πρέπει να μπορέσει να λειτουργήσει σε φάσεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στους πληθυσμούς. Θα πρέπει η Επιτροπή να προχωρήσει λοιπόν σε αξιοποίηση των εμπειριών των εθελοντών, αναγνωρίζοντας όπως είπα τις ικανότητες τις οποίες έχουν αποκτήσει στον επαγγελματικό τους και κοινωνικό χώρο η ιδέα των Ευρωπαίων εθελοντών είναι μια εξαιρετική ιδέα. Είναι μια ιδέα που προσφέρει ε, στην ιδέα της Ευρώπης τους πληθυσμούς μας. Ξέρω ότι δημοσιονομικά θα έχουμε προβλήματα και αύριο θα το συζητήσουμε αυτό με την Ιρλανδική Προεδρία. Μια παρένθεση επιπλέον σχετικά με το κοινό νομικό καθεστώς. Είναι απαραίτητο να βρεθεί μια λύση στον τομέα αυτό γιατί ε, η έλλειψη λύσης ε, θα μεγενθύνει τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νιούτον Ντάουν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Ζητώ συγγνώμη, ήρθα λίγο καθυστερημένα. Συνεπώς αν πω κάτι λάθος, συγχωρέστε με. Δεν είχα καταλάβει ότι είχε αλλάξει προτεραιότητα στην ημερησία διάταξη. Εγώ παρακολούθησα την προπαρασκευή των εθελοντών και ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα σχόλιά τους. Είναι εξαιρετικά καλή ιδέα αυτό το πρόγραμμα και ελπίζω να απογευθεί και να πετάξει τέλεια. Αλλά έχω τρεις μικρές ερωτήσεις. Η πρώτη με την δημοσιονομική λιτότητα και τη μάχη με τα κράτη-μέλη για οποιαδήποτε αύξηση του ετήσιου προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Γνωρίζει η Επιτροπή κατά πόσο είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν χρήματα για το πρόγραμμα ή αν θα χρειαστεί να κυρωθούν άλλα προγράμματα ώστε να βρεθούν χρήματα γι' αυτό. Είναι ένα ζήτημα αυτό του προπολογισμού. Σοβαρό και δύο άλλα μικρά σημεία που προκύπτουν από τις προπαρασκευαστικές ε, συναντήσεις της εκθέσης των εθελοντών. Το πρόβλημα, το ζήτημα των γλωσσών. Δεν καταλάβαιναν όλοι ο ένας τον άλλο. Δεν είχαν κάποια κοινή γλώσσα. Το οποίο είναι κατανοητό. Σε αυτήν εδώ την Επιτροπή έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Αλλά είμαστε τυχεροί. Έχουμε τους δερμηνείς που μας βοηθούν. Έχει σκεφτεί κανεί ε, για το τι θα κάνουμε με αυτή την πολυγλωσία των διαφόρων εθελοντών και πώ μπορούν αυτού να συνεργαστούν μεταξύ του. Και τέλος, όσον αφορά τις αποζημιώσεις, τα χρήματα που κερδίζουν οι εθελοντές φαντάζομαι ότι τους πληρώνετε σε διαφορετικό επίπεδο ανάλογα με τη χώρα στην οποία πηγαίνουν και πρέπει να είναι αρκετά σύνθετο αυτό το ζήτημα. Φαντάζομαι ότι μελετάτε και κάποιο μηχανισμό για να επιληθεί αυτό. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ. Κυρία Θεοχάρους, έχετε το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική παρουσίαση. Και έχω ένα σχόλιο. Ουσιαστικά ήταν ερώτηση στην αρχή, αλλά... Μετά από τα όσα είπε ο συνάδελφος, είναι περισσότερο σχόλιο. Όταν μιλάμε για αποζημιώσεις μισθούς ε, για τους εθελοντές, τότε δεν είναι εθελοντές. Αν πρόκειται να προσλαμβάνουμε εμπειρογνώμονες εργαζόμενους επιτόπου δεν είναι σωστό να μιλάμε για εθελοντές, ούτε για εθελοντισμό. Ευχαριστώ. Merci. La parole est à Monsieur Cortes Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Κόρτες Λάστρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον υπεύθυνο για αυτή την παρουσίαση που ήταν τόσο ενδιαφέρουσα. Εξαιρετική δουλειά είναι αυτή που έγινε. Και όχι μόνο κάνουμε λόγο για πρόσθετη ευρωπαϊκή αξία όπως ανέφερε, αλλά δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την λέξη πρόσθετη αξία, αλλά αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντανακλώνται. Γι' αυτό το πρόγραμμα και σχέδιο που έχουμε στα χέρια μας θα προσεγγίσει περισσότερο τους πολίτες σε αυτή τη συνεργασία και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες ανεξάρτητα από το αν συμμετέχουν ή όχι σε αυτά τα προγράμματα συνεργασίας θα αισθάνονται ότι κάποιος πολύ κοντινός σε αυτούς, ένας πολίτης νέος ή όχι θα μπορεί να συνεργάζεται και να εντάσσεται σε αυτές τις τόσο σημαντικές αξίες δηλαδή αλληλεγγύη. Από αυτό, περί αυτού πρόκειται. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα φυσικά να συγχαρώ, να συγχαρώ τον υπεύθυνο και να κάνω δύο ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση έκανε λόγο και είπε θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το βλέπουμε να αναπτύσσεται στο διαδίκτυο και στο δίκτυο αυτό μέσω των εργασιών του έργου των εθελοντών. Ερώτηση, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πώς μπορούμε εμείς να συνεισφέρουμε, να αντλήσουμε αυτές τις γνώσεις και αυτή την πείρα στο δίκτυο, στο δίκτυο αυτό με τους υπόλοιπους τους εθελοντές που μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θετικό για την ευρωπαϊκή συνεργασία αυτό το, αυτή, αυτό το εγχείρημα και ε, σε ένα ε, ίσονος ε, θέμα την Κεντρική Αμερική, δεν κάνω λόγο για τη Λατινική Αμερική, για την Κεντρική Αμερική που είναι συγκεκριμένη περιοχή με πολύ έντονα οξέα προβλήματα. Θα μπορούσε εκεί κάτι να γίνει μέσω αυτών των ε, οργανώσεων, να υπάρχει για παράδειγμα κάποιο πρόγραμμα, κάποιο σχέδιο για, το, ε, για την συνεργασία, μια και έχουν προβλήματα όλο και περισσότερο έντονα για συγκεκριμένα θέματα που δεν έχουμε χρόνο τώρα να επισέλθουμε σε αυτά. Θα έπρεπε να υπάρξει λοιπόν μια τέτοια δυνατότητα να μπορούν να συνεργαστούν τέτοιου είδους εθελοντές εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια και πάλι. Κύριος Νόισερ θα λάβει τον λόγο παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια και από πλευράς μου. Όμως πρέπει σε αυτά τα συγχαρητήρια και την Επίτροπο Γεωργίευα να συμμετάσχουμε, να εντάξουμε. Πώς επίτροπος παρουσιάστηκε στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ώστε αυτή η εθελοντική υπηρεσία να είναι ένα από τα κύρια θέματα που την ενδιέφεραν. Και τώρα βρίσκεται υπό εξέλιξη αυτό και είναι εξαιρετικό. Και η παρουσίαση ήταν διεξοδική και πολύ καλή. Θα έλεγα η ευρωπαϊκή πρόσθετη αξία που απορρέει θα πρέπει να βρίσκεται σε ισόρροπο λόγο, σε ισόρροπη αναλογία με την αποτελεσματικότητα αυτής της υπηρεσίας. Τι γίνεται, υπάρχουν δυνατότητες αυτός ο ισολογισμός μεταξύ αποτελεσματικότητας και ευρωπαϊκής πρόσθετης αξίας στα επιμέρους αυτά σχέδια να παρουσιάζεται πιο καλά και να έχει ε, πιο ανάγλυφη αξία. Και είπατε ότι υπάρχει online διαδικτυακά μια τέτοια κατάρτιση. Διαδικτυακά μόνο πρόσθετη εκπαίδευση ή κατάρτιση μπορεί να είναι στην κανονική εκπαίδευση ή κατάρτιση γιατί με μια καθαρή online εκπαίδευση ή κατάρτιση θα είχαμε πολλές επιφυλάξεις. Τελευταία παρατήρηση, corporate identity, δηλαδή ε, στη συλλογική αυτή ένταξη ή παρουσίαση είναι πολύ σημαντικό αυτό. Χρειαζόμαστε μηνύματα επιτυχή από την Ευρώπη προς τα έξω. Δεν μπορεί να είναι μια εθελοντική υπηρεσία που μετά θα, θα υποβαθμίζεται εθνικά μέσω άλλων ε, συνιστοσών. Θέλουμε να υπάρχει αυτή η κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο ξανά στον Μάρκο Χέλτ για να απαντήσει. Κύριε Χέλτ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω κάποιες από αυτές, αλλά θα αφήσω φυσικά και του συναδέλφους μου που ακολουθούν τη συναντήση που να απαντήσουν. Θα ξεκινήσω από τα ζητήματα που αφορούν την κατάρτιση. Ακούστηκαν πολλές τέτοιες ερωτήσεις. Αυτό σε αυτό το σημείο δεν συμφωνούμε απόλυτα με τους ΜΚΟ. Στον κανονισμό έχουμε ένα πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα αναπτύξει η Κομισιόν. Αλλά τι εννοώ με αυτό. Θα βασιστούμε σε ό,τι ήδη υπάρχει. Δεν θα επινοήσουμε εμείς ε, εκπαιδευτικά προγράμματα που ήδη υπάρχουν. Παρατηρήσαμε όμως ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προτείνουν οι διάφοροι οργανισμοί είναι αλληλοσυμπληρωματικά. Κάποια έχουν πιο ισχυρά σημεία από άλλα και αυτό που θέλουμε εμείς είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο θα καταλήξουμε να λαμβάνει υπόψη ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να φοβάται ο τομέας ούτε η μήκα. Ο μικρόν δεν πρόκειται να επινοήσουμε κάτι καινούριο. Θα γίνουν όλα αυτά σε στενή συνεργασία. Αυτή τη στιγμή ε, οριστικοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα κάνουμε μια πρόσκληση υποβολής προσφορών, στην οποία μπορούν να απαντήσουν ένας ή περισσότεροι οργανισμοί για την διεξαγωγή του εκπαίδευση. Δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα οι ίδιοι οργανισμοί, διότι είδαμε στα πιλωτικά προγράμματα ότι σκόπιμο είναι να έχουμε εθελοντές από διαφορετικά προγράμματα μαζί, να εκπαιδεύονται μαζί και να αναπτύσσονται στη συνέχεια από τους οργανισμούς τους. Να αποστέλλονται από τους οργανισμούς τους. Δεν είναι αυτόματο λοιπόν το σύστημα. Όπως προείπα, το πρόγραμμα αυτό θα βασιστεί σε ότι ήδη υπάρχει και ελπίζουμε ότι θα είναι λίγο πιο πλήρες από τα επιμέρους προγράμματα των διαφορών μικαπόμικρων. Φυσικά δεν θα είναι μόνο ένα πρόγραμμα online στο διαδίκτυο. Η εκπαίδευση στο διαδίκτυο δεν είναι παρά ένα κομμάτι. Μιλάμε για blended learning, μεικτή εκμάθηση, δηλαδή ένα μείγμα μεταξύ επιτόπου ε, κατάρτισης αλλά και κατάρτιση προπαρασκευή online. Δεν θα είναι λοιπόν ποτέ αποκλειστικά και μόνο στο διαδίκτυο. Συμφωνούμε σε αυτό. Για το ζήτημα των γλωσσών. Ναι, πράγματι προέκυψε αυτό το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να διαβρούμε διάφορες λύσεις. Δεν έχω λοιπόν να σας δώσω κάποια συγκεκριμένη απάντηση, έτοιμη απάντηση, γι' αυτό μία επιλογή θα μπορούσε να είναι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στον τρόπο υλοποίηση του προγράμματος να υπάρχουν διαφορετικές γλωσσικές εκδόσεις της εκπαίδευσης, δηλαδή να προσφέρεται εκπαίδευση στα αγγλικά, στα γαλλικά ή στα ισπανικά αυτή είναι μία από τις επιλογές. Αλλά όπως σας είπα δεν έχουμε απάντηση έτοιμη. Από την άλλη, οι διαπολιτισμικές εμπειρίες ε, στα πιλωτικά προγράμματα που είχαμε ήδη οφείλονταν ακριβώς στο γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν μιλούσαν τις ίδιες γλώσσες. Δηλαδή το να συγκεντρώνουμε ανθρώπους από διαφορετικά περιβάλλοντα και να τους οθούμε να βρουν μια κοινή γλώσσα να βγουν από τη γλωσσική του ομάδα και αυτό μπορεί να προσφέρει θέμενη αξία στο πρόγραμμα. Όπως είπα, είναι μια διαδικασία την οποία ακόμα μελετάμε για να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το ζήτημα τώρα του εθελοντισμού είναι σημαντικό. Φυσικά δεν πρόκειται να καταβάλουμε μισθούς. Παραμένουν εθελοντές αυτοί οι άνθρωποι, αλλά πρέπει να μπορούν και να ζήσουν. Μιλάμε λοιπόν για αποζημιώσεις που επιτρέπουν στους ανθρώπους να αγοράζουν τρόφιμα, να επιβιώνουν και η αρχή που εφαρμόζουμε είναι ότι οι εθελοντές αυτοί δεν πρέπει να πλήρωνουν από την τσέπη τους τον εθελοντισμό που προσφέρουν. Δηλαδή κατά βάση από την αρχή ως το τέλος του προγράμματος δεν θα πρέπει να βάζουν αυτοί χρήματα ούτε να κερδίζουν. Αυτή είναι η αρχή που εφαρμόζουμε εμείς. Μηδέν κέρδος δηλαδή αθρηστικά για κάθε εθελοντή. Εκεί λοιπόν υπάρχει διαφορά μεταξύ εθελοντή και μισθωτού. Τώρα, όσον αφορά τη δημοσιονομική λιτότητα και κατά πόσο είμαστε βέβαιοι ότι ο προπολογισμό θα είναι επαρκή, θα απαντήσει η Τζούλια σε λίγο. Όσον αφορά τη δικτύωση των εθελοντών, μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Στα διάφορα πιλωτικά προγράμματα παρατηρήσαμε ότι χρησιμοποιούνται διαφορετικά μοντέλα Κάθε πιλωτικό πρόγραμμα έχει κάποιον online χώρο συνεργασίας όπου αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι εθελοντές, ανταλλάσσουν πληροφορίες ε, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και διάφορες άλλες πληροφορίες. Επίσης ε, είχαμε και άλλες εμπειρίες στο δίκτυο Νόχα ε, φοιτητές πανεπιστημίων που ανήκαν ε, στο δίκτυο φοιτητών και μετά στο δίκτυο αποφύτων, με αλληλοϊποστήριξη. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί τρόποι όπως έχουμε παρατηρήσει τα πιλωτικά προγράμματα και κοιτάμε να δούμε τι θα υλοποιήσουμε. Ένα κομμάτι από αυτό θα είναι το online πρόγραμμα εθελοντισμού, αλλά ένα άλλο κομμάτι επίσης θα είναι και ένα δημόσιο φόρουμ όπου όλοι θα μπορούν να ενημερώνονται να διαβάζουν ιστολόγια, να διαβάζουν ιστορίες, εμπειρίες από την επιτόπου δράση και εξετάζουμε εμείς το πώς ακριβώς θα αναπτύξουμε αυτού του είδους το δίκτυο. Ήθελα να πω και κάτι για την Κεντρική Αμερική και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους ε, για να βεβαιωθούμε ότι θα απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Στην Κεντρική Αμερική ξέρω ότι υπάρχει μία χώρα, αλλά πρέπει, δεν θυμάμαι ποια, όπου το πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού πολιτική Προστασία του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού έστειλε κόσμο στην Κολομβία και σε μια κεντροαμερικανική χώρα που δεν θυμάμαι ποια είναι. Υπάρχουν δηλαδή χώρε που καλύπτονται ήδη, αλλά ακόμα βρισκόμαστε σε πιλωτική φάση. Θα ακολουθήσουν και άλλα και δίνω τώρα το λόγο στην Τζούλια για να απαντήσει τα υπόλοιπα. Thank you very much. Um, Julie Stewart David uh, from the Είμαι αναπληρώτρια διευθύντρια της διεύθυνσης από την οποία προέρχεται και ο Μάρκ. Θα ήθελα να πω ότι πέρα από το θέμα της εμπιστοσύνης που θέσατε για τον προϋπολογισμό, είναι δύσκολη απάντηση. Εμείς είμαστε πεπισμένοι για το καλό της πρότασής μας. Έχουμε κάνει μια καλή ανάλυση κόστους και ωφέλους 239 εκατομμύρια για τα 7 χρόνια για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι σε διαφορετική γραμμή από αυτόν ο οποίος προτείνεται για την ανθρωπιστική βοήθεια που γίνεται αντικείμενο διαχείρισης γενικότερα από την Επιτροπή. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι υπάρχει κάποια ανησυχία, και αυτό δεν εκπλήσει κανέναν από τα κράτη-μέλη, για μια νέα πρωτοβουλία και το κόστος αυτής της νέας πρωτοβουλίας σε μια δύσκολη φάση. Αυτό αντικατοπτρίζεται όμως από μια γενικότερη μορφή στήριξης από πλευράς άλλων κρατών μελών. Στην παρούσα φάση θα ήθελα να πω ότι εμείς κάνουμε αυτή την δημοσιονομική πρόταση σε ένα επίπεδο την οποία θεωρούμε ρεαλιστική αλλά και φιλόδοξη. Η Επιτροπή δεν θα ήθελε να μειωθεί ιδιαίτερα το μέγεθος των φιλοδοξιών μας. Ένα από τα πιο ακριβά στοιχεία είναι ακριβώς η ανάπτυξη αυτών των εθελοντών. Έχουν γίνει κάποιες προτάσεις ότι στον τομέα αυτό θα μπορούσαμε ίσως να μην κάνουμε αναφορά στην πρόταση. Αυτό δεν είναι σωστό. Εμείς θεωρούμε ότι το θέμα αυτό είναι τμήμα του προγράμματος. Δεν μπορώ να φανώ προφήτης, αν έχουμε να κάνουμε με έναν μειωμένο προϋπολογισμό, σε ένα κάποιο επίπεδο θα εργαστούμε μέσα στο μειωμένο προϋπολογισμό. Αν το επίπεδο είναι πολύ πιο χαμηλό, τότε θα πρέπει να τα επανεξετάσουμε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην κυρία Στρίφλερ για να κλείσει τη συζήτηση. Κοιτάξτε, δεν έχω και εγώ τίποτα άλλο να προσθέσω. Ήταν πλήρης η παρουσίαση έχουν υπάρξει κάποια στοιχεία επί των οποίων θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος, εντοπίστηκαν, αλλά νομίζω ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό πρόγραμμα, δεν το λέω για την δική μου η έκθεση. Ξέρουμε τι λέει η εμπειρία μας επί υπάρχει μια καταστροφή, ο αριθμός των ανθρώπων που θέλουν να προσφερθούν εθελοντικά, είτε είναι νέοι είτε και λιγότερο νέοι, νέοι, ναι, γενικά συνταξιούχοι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή και να κάνουμε μια εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε τώρα. Έπρεπε να είναι κανονικά εδώ ο κύριος Κάσμαν, ο οποίος θα μας παρουσίασε ε, την δική του έκθεση, αλλά το τρένο του θα καθυστερήσει, θα φτάσει μετά τις 5 και γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω να πάμε τώρα στο σημείο 12 πριν το 11. Βοήθεια για την ανάπτυξη λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πόσιμου ύδατος και των υπηρεσιών καθαρισμού των υδάτων και των λιμάτων στις υποσαχαρικές χώρες. Έχουμε και μια έκθεση επίσης της, του ελεγκτικού συνεδρίου στα πλαίσια της απαλλαγής για το 2011 σχετικά με τη βοήθεια για την ανάπτυξη, για το πόσιμο είδωρ και την επεξεργασία των λιμάτων. Καλωσορίζω εδώ το μέλος του συνεδρίου, το υπεύθυνο, για το συγκεκριμένο θέμα, David Μπόστοκ γνωμοδότης της Επιτροπής μας προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού που είναι επί της ουσίας υπεύθυνη είναι η κυρία Ζαμπόρσκα η οποία είναι μαζί μας σήμερα. Θα ξεκινήσω δίδοντας το λόγο στον κύριο Μπόστοκ ε, του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να μας παρουσιάσει την δική του ε, έκθεση. Ο έλεγχος αυτός αφορά ένα σημαντικό κομμάτι της ε, ε, υπερατλαντικής βοήθειας, θα έλεγα, ή μάλλον της βοήθειας προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο λόγο λοιπόν ε, όλο αυτό ζητήσαμε τα έργα αρρωγής για πόσιμο νερό και υποδομές αποχέτευσης να οδηγούν σε αϊφόρα αποτελέσματα κατά πόσο λοιπόν είναι βιώσιμα τα αποτελέσματα και κατά πόσο η Κομισιόν έκανε ό,τι μπορούσε και ό,τι έπρεπε να κάνει ώστε να μπορέσει να επιτύχει βιώσιμα αποτελέσματα. Πώς εκτιλήσετε το έργο αυτό. Αξιολογούμε την επιτυχία 23 έργων στην Αγγόλα, στον Πενίν, στην Μπουρκίνα Φάσο, στην Κάνα, στην Ιγυρία και στην Τανζανία. Ο οικονομικός έλεγχος εξετάζει αρχεία και εκθέσεις σε σχέση με τα προγράμματα, για παράδειγμα εκθέσεις παρακολούθησης και εξολόγησης από την Κομισιόν και για την Κομισιόν. Επίσης, οι οικονομικοί ελεγκτές επισκέφθηκαν τρεις από τις ε, σχετικές χώρες, την ε, Μπουρκιναφάσο, Νιγηρία και Τανζανία. Τι ανακαλύψαμε. Για ανάμεικτη εικόνα. Πρώτον, γενικώ και εγκατασταθεί εξοπλισμός με κάποιες προσαρμογές για τις τοπικές συνθήκες και ήταν σε λειτουργική κατάσταση. Δεύτερον, ωστόσο, οι ανάγκες των δικαιούχων, όπως ορίζονται στα προγράμματα, ε, πληρούνταν σαφώς μόνο σε δύο περιπτώσεις και με κάποιες ελλείψεις σε επιπλέον έξι περιπτώσεις. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις υπήρχαν πολύ σοβαρότερες ελλείψεις. Τρίτον, βιωσιμότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι μπορούσαμε να δώσουμε καλή βαθμολογία στα προγράμματα όσον αφορά την τεχνική βιωσιμότητα. Χρησιμοποιήθηκε στάνταρ, τεχνολογία και τοπικά διαθέσιμα υλικά. Ωστόσο αυτό που ήταν λιγότερο ικανοποιητικό ήταν η οικονομική βιωσιμότητα και η θεσμική βιωσιμότητα. Όπως ονομάζονται τα έργα παροχής πόσιμου νερού και αποχέτευσεων θα μπορούσαν να παρέχουν συνεχή ωφέλη εάν παρήχαν επαρκή έσοδα ώστε να καλύπτονται τα τρέχοντα έξοδα, η συντήρηση και επισκευές ρουτίνες και εφόσον αυτό είναι δυνατόν να γίνεται ικανοποιητικά. Προσπάθησε λοιπόν το ελεκτικό συνεδρίο να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα τέτοιων εσόδων από δασμούς, από περαιτέρω πληρωμές ή από άλλου τύπου έσοδα και κατά πόσο είναι δυνατή η ικανοποιητική λειτουργία. Και διαπιστώσαμε τα εξή. Σε τέσσερα έργα είχαν δημιουργηθεί δασμοί έτσι ώστε να καλύπτονται τα έξοδα λειτουργία σε τρει περιπτώσει. είχαν λάβει μέσα οι τοπικέ αρχέ, ώστε να υποστήριζονται τα έργα όπω ήταν απαραίτητο παρότι δεν τηρούσαν αυτέ τι δεσμεύσει. Αλλού δεν υπήρχαν καν τέτοιε δεσμεύσει και σε σημαντικό αριθμό προγραμμάτων είδαμε προβλήματα όσον αφορά τη θεσμική βιωσιμότητα, δηλαδή έλλειψη τεχνικών ικανοτήτων, η έλλειψη οικειοποίησης και πλήρους ανάληψη ευθύνης για έργα. Το ελεγκτικό συνέδριο είναι ένας οργανισμός οικονομικού ελέγχου και όχι προβλέψεων. Δεν μπορούμε λοιπόν να προβλέψουμε το μέλλον. Θεωρήσαμε όμω ότι ήταν απαραίτητο να συμπεράνουμε, όπω θα δείτε στη σύνοψη τη έκθεσης, ότι στην πλειοψηφία αυτών των έργων τα αποτελέσματα και τα ωφέλη δεν θα συνεχίσουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, εκτό εάν διασφαλιστεί, διασφαλιστούν μη δεσμολογικά έσοδα ή λόγω θεσμικών ελλείψεων. Και εδώ καταλήγουμε στο τελευταίο κομμάτι των διαπιστώσεων του ελεκτικού συνεδρίου, ο τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την υποστήριξη για αυτά τα έργα η Κομισιόν. Η Κομισιόν, λοιπόν, ανέπτυξε πολύ σωστά διευθετήσεις για διαχείριση έργων που ε, βοήθησαν τη δυνατότητα βιωσιμότητας των έργων. Στα χαρτιά όλα φαίνονται μια χαρά. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώσαμε ότι πρακτικά η διαχείριση έργων δεν επιβίωσε όπως θα επιβίωνε θεωρητικά σημαντικές ελλείψεις ε, στον ορισμό τεχνικών και οικονομικών στόχων, οι ασαφείς στόχοι, οι δείκτες πρόοδου. Ειδικότερα οι ελεγκτές ε, βρήκαν ελάχιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε αντιμετωπιστεί το ζήτημα δημιουργίας κονδυλίων για την κάλυψη τρεχόντων δαπανών έργων. Τι πρότεινε τελικά το ελεγκτικό συνέδριο. Οι συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου απορρέουν από τις παρατηρήσεις μας. Μετά από τους ελέγχους, η Κομισιόν θα πρέπει να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται σωστά οι διαδικασίες της και θα πρέπει να μεριμνά ιδιαίτερα ώστε να υπάρχει εύλογη προοπτική μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης υποστήριξης των προγραμμάτων όπως απαιτείται. Αυτά ήθελα να σας πω εισαγωγικά. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Σαμπόσκα για την άποψή της. Um, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ που μου αναθέσατε αυτή τη γνωμοδότηση. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να ασχολιάσει κανείς μια ειδική έκθεση ε, του ελεγκτικού συνεδρίου που ασκεί κριτική στην κοινοτική πολιτική στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Η ειδική έκθεση παρίθμου 13 του 2012 έχει σαν βασικό στόχο το μη στον τομέα του πόσιμου ύδατος και της επεξεργασίας των λιμάτων στην υποσαχαρική Αφρική. Είπα ότι η προσπάθεια αυτή θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δύσκολη γιατί θα πρέπει να βρει κανείς μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στο θέμα του σεβασμού της χρήσης των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων και την χρήση των πόρων που είναι διαθέσιμοι για την επιβίωση των συμπολιτών μας στην Αφρική. Εδώ τίθεται και το θέμα της σκιάς, έλεγα πάνω σε όλα αυτά, της πολιτικής ορθότητας. Στην πραγματικότητα η κατάσταση ε, στον τομέα των υδάτων στον κόσμο είναι πολύ ανησυχητική και γι' αυτό και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών διόρισε ένα ειδικό εισηγητή, την κυρία Κάτεριν Αλμπουκέρκ, υπεύθυνη για την επεξεργασία των ε, υδάτων και το πόσιμο είδωρ στα πλαίσια των στόχων της νέας χιλιετίας. Παρ' όλα αυτά, το είδωρ και η επεξεργασία των λιμάτων όπως και τα τρόφιμα άλλωστε είναι εγκάρσιες και θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την επίτευξη όλων των στόχων της χιλιετίας για τους πολίτες του κόσμου αυτού ανεξαρτήτως γενεάς. Γι' αυτό και η σημασία του ύδατος στις διεθνείς σχέσεις και στην πολιτική συνεργασία για την ανάπτυξη. Σας προτείνω λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας ότι θα πρέπει εμείς να ασχοληθούμε ειδικά με τον σημαντικό αυτό παράγοντα της ανάπτυξης μέσω της επεξεργασίας μιας νομοθετικής εκθέσεως της οποίας θα προηγηθεί μια δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή των πρέσβειων των χωρών της υποσαχαρικής Αφρικής. Η παρούσα έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αφορά την αξιολόγηση των επιδόσεων της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της προμήθειας πόσιμου ύδατος και της επεξεργασίας των λιμάτων στην Ποσαχαρική Αφρική. Θέλει το, το ελεγκτικό συνέδριο να δει αν πράγματι πετυχαίνουμε τους στόχους μας της παρέμβασης αυτής. Όπως είπε ο κύριος Μπόστοκ και τον ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση της έκθεσής του, το ελεγκτικό συνέδριο προχώρησε στον έλεγχο 23 προγραμμάτων σε 6 χώρες. Αγγόλα, Μπενέ, Μπουρκίνα Φάσο, Γκάνα, Νιγερία, Τανζανία. Η οικονομική εμπλοκή της Ένωσης ανέρχεται σε 219 εκατομμύρια ευρώ ανάμεσα στο 11 και στο 10 για το σύνολο των 46 χωρών η Επιτροπή έχει επενδύσει άνω των 2 δις ευρώ. Κατά συνέπεια η ειδική έκθεση που έχουμε μπροστά μας του ελεγκτικού συνεδρίου αναφέρεται στο 1 τέταρτο των προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από την Ένωση ελέγχοντας την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών μας και των πιθανών συνεπειών τους. Τις βασικές παρατηρήσεις δεν θα τις επαναλάβω γιατί τις παρουσίασε ο κύριος Μπόστοκ. Να προσθέσω όμως εδώ ότι το συνέδριο συνιστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πολλούς τομείς να χρησιμοποιήσει καλύτερα τις υπάρχουσες διαδικασίες για να μεγιστοποιήσει τα πλεονεκτήματα των πιστώσεων αυτών στην ζώνη αυτή και για τον τομέα στον οποίο προαναφέρθηκα. Ανεξαρτήτως του θέματος ε, του ύδατος, είχα ήδη πει κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής διαδικασίας ότι τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλευση χρημάτων να ληφθούν υπόψη και από τους οργανισμούς τους οποίους έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τους νόμιμους εκπροσώπους των τοπικών πληθυσμών οι οποίοι θα μας έλεγαν αν οι χρηματοδοτήσεις ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Θα βρείτε όλες τις παρατηρήσεις μου λοιπόν στο σχέδιο γνωμοδότησης και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τη γραμματεία της Επιτροπής μας για την προσπάθειά της και την ευελιξία της και τις σωστές της προτάσεις. Οι παρατηρήσεις σας ήσαν καλοδεχούμενες και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ζαμπόσκα. Το λόγο έχει ο κύριος Γκουερέρο Σάλλον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τον εκπρόσωπο που μας διατύπωσε και παρουσίασε αυτή την πείρα το έργο το οποίο υλοποιήθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο όσον αφορά την υδροδότηση ή την παρακολούθηση και συνοδευτική παρακολούθηση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υδροδότηση και το καθαρό πόσιμο νερό για τις υπο... μεσημβρινές ε, υποσαχάριες αφρικανικές χώρες. Κάποιες ερωτήσεις θα διατυπώσω στο τέλος της παρέμβασής μου. Όμως πρώτα θα ήθελα να κάνω αναφορά σε κάτι που πιστεύω ότι όλους μας απασχολεί και το θυμόμαστε. Είναι η στρατηγική σημασία που έχει η πρόσβαση στο νερό. Όχι μόνο για την καταπολέμηση της ε, πείνας, μια και η έλλειψη νερού βρίσκεται ως αίτιο στην αρχή όλων των λιμών που μαστίζουν την Αφρική και άλλες περιοχές του κόσμου, ιδιαίτερα την υποσαχάρη Αφρική, αλλά και από την άλλη πλευρά επειδή οι σειράξει και οι αντιπαραθέσεις για το νερό βρίσκονται στα αίτια πολλών σειράξεων που οδηγούν στο να χάσουν τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι, καμιά φορά εκατομμύρια άνθρωποι. Και γι' αυτό λοιπόν όλα εκείνα που μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσουμε, να παράσχουμε και να εγγυηθούμε την πρόσβαση στο νερό σε αυτό το τμήμα αυτής της Υπήρου είναι μια δράση που στοχεύει την καταπολέμηση της ε, πείνας και μια δράση που θα διατηρεί την ειρήνη ή θα οδηγεί προληπτικά στην αποφυγή σειράξεων. Ωστόσο από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε από τις αξιολογήσεις που κάνουμε ότι η πρόσβαση στο νερό είναι ένας από τους κύριους στόχους της χιλιετίας που πόρο απέχουμε από το να έχουμε υλοποιήσει και γι' αυτό είναι Μία από τις πτυχές επί των οποίων αν θέλουμε να προσεγγίσουμε το 2015 αυτά που δεσμευθήκαμε να προσεγγίσουμε το 2000 πρέπει ακόμα περισσότερες προσπάθειες να κάνουμε. Περισσότερες επιπρόσθετες ακόμη προσπάθειες. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου καταδεικνύει σαφώς μέχρι ποιο σημείο είναι δύσκολο στην για την Ευρωπαϊκή Ένωση η υλοποίηση και εφαρμογή των συγκεκριμένων εξειδικεμένων προγραμμάτων για το νερό, την παροχή νερού και καθαρού πόσιμου ύδατος και μέχρι ποιού βαθμού μπορεί να βελτιωθεί η δουλειά μας που υφίσταται ε, περιορισμούς ε, από αυτό το έργο, ιδιαίτερα όσον αφορά αυτή την πτυχή της αξιολόγησης. Έχουμε συνειδητοποιήσει, απόλυτα έχω συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες του να προχωρήσει αυτό το έργο από πλευρά μα. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιοι μηχανισμοί είναι εκείνοι που χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να διασφαλιστεί η χνηλασιμότητα. Να βρούμε δηλαδή την ανείχνευση του τι κάνει η επίσημη βοήθεια για την ανάπτυξη σε σχέση με το νερό συγκεκριμένα. Θα ήθελα να ξέρω στο πολιτικό διάλογο που κάνουμε και διαμορφώνουμε και υλοποιούμε με τους εταίρους μας στην ε, Ήπειρο αυτή, αν έχει συμπεριληφθεί συστηματικά έχουν συμπεριληφθεί τα θέματα που αφορούν το νερό και την, τον καθαρισμό, την, ε, το πόσιμο νερό. Και θέλω να πω, όταν πριν ανέφερα ότι είναι θεμελιώδους σημασίας το νερό για την καταπολέμηση της πείνας και για τη διασφάλιση της ειρήνης είναι αποφασιστικός παράγοντας, παράγοντας για την κατάκτηση της υγείας. Έχει πολλές συνιστώσεις και πτυχές η υγεία και τη μητρότητα και την επιβίωση των παιδιών, των βρεφών. Δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς ε, τους στόχους της χιλιετίας χωρίς να υπάρχει παροχή νερού σε αυτές τις κοινότητες που δεν έχουν στη διάθεσή τους το νερό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκέρενς, έχετε το λόγο. merci, madame la... Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μου κάνει έκπληξη αρνητική χρειά της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου όσον αφορά την πρόσβαση σε πόσιμο νερό και τα έργα που σχετίζονται με την υδροδότηση και την αποχέτευση στην υποσαχάρη Αφρική. Είναι ιδιαίτερα σκληρό το ελεγκτικό συνέδριο όσον αφορά δύο πτυχές στην ικανότητα οικειοποίηση των προγραμμάτων και όσον αφορά τη βιωσιμότητα που φαίνεται να είναι αρκετά ανεπαρκής. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία που αναφέρθηκαν. Για μένα η οικειοποίηση ουσιαστικά αποτελεί σημαντική στιγμή στην ιστορία, στον κύκλο ενός έργου. Η επίσημη οικειοποίηση είναι η στιγμή κατά την οποία ή μάλλον από την οποία ο δικαιούχος γίνεται ιδιοκτήτης του προγραμματός του και μετά ακολουθεί η ανάληψη ευθύνη από τον ιδιοκτήτη αυτού του έργου. Αυτό που μου κάνει έκπληξη λοιπόν είναι το γεγονός ότι πρακτικά η μεγάλη πλειοψηφία προγραμμάτων φαίνεται να είναι ανεπαρκή για τους ε, υπεύθυνου αξιολόγηση του ελεκτικού συνεδρίου. Έχω κάποιες ερωτήσεις και μετά θα κάνω κάποιο σχόλιο. Το πρώτο ερώτημα είναι, έχετε διαπιστώσει ότι στις χώρες όπου τρέχουν προγράμματα τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά από τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε χώρες όπου παρέχει δημοσιονομική αρρωγή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσατε να μας πείτε τη δική σας άποψη, τη δική σας εκτίμηση για αυτή την πτυχή των πραγμάτων. Μου φαίνεται σημαντικό αυτό. Αναρωτιέμαι επίσης ε, κατά πόσο στις ε, χώρες που λαμβάνουν ε, δημοσιονομική αρρωγή, όπου η Κομισιόν ε, κυρίως επιμένει στη βελτίωση της διακυβέρνησης, εάν και εκεί απαντάτε αυτά τα προβλήματα. Διότι η δημοσιονομική στήριξη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο επίπεδο ικανότητας διαχείρισης του προπολογισμού από τη χώρα δικαιούχο. Δεύτερον, έχετε διαπιστώσει δυσκολίες ε, σε επίπεδο τοπικής διακυβέρνησης. Εκεί έχετε περισσότερα προβλήματα, διότι νομίζω τα ε, περισσότερα προβλήματα πρόσβασης στο νερό, στα ύδατα, ε, τη χάνουν διαχείριση σε επίπεδο Δήμου. Οι Δήμοι λοιπόν εκεί οι άλλοι συμμετέχοντες ποιοι είναι αυτοί που ασχολούνται με αυτά και Τέλος, μια ερώτηση όχι απαραίτητα προς το ελεγκτικό συνέδριο, μια ερώτηση προς την Κομισιόν και προς εμάς τους ίδιους πολιτικό συμπέρασμα. Έχετε κάποιο καταμερισμό εργασιών στο πλαίσιο της ατζέντα για την ανάπτυξη. Εμείς συμφωνούμε στο πλαίσιο αυτό, λέει η Κομισιόν, ότι δεν θέλει να υλοποιεί υπερβολικά πολλά προγράμματα στην ίδια χώρα, θέλει να περιορίζεται σε τρεις τομείς το πολύ. Μήπω καλό θα ήταν να ειστεστεί περισσότερο η Κομισιόν στη βελτίωση της διακυβέρνησης αντί να συνεχίζει να υλοποιεί τεχνικά προγράμματα διότι όταν υλοποιεί κανείς τεχνικά προγράμματα και ταυτόχρονα εμπλέκεται σε προγράμματα βελτίωση της διακυβέρνησης εκεί εμπλέκεται κανείς, δεν θα έλεγα σε διένεξη συμφερόντων, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να είστε δικαστής και αναγόμενος ταυτόχρονα. Έχετε ας πούμε κάποια έργα που επιτυχάνουν σε κάποια αφρικανική χώρα και ταυτόχρονα έχετε και κάποια ευθύνη βελτίωσης της διακυβέρνησης. Δεν είμαι βέβαιος. Καθώς τα μέσα που διαθέτουμε είναι ούτως ή άλλως περιορισμένα, πώς θα ήταν καλύτερο να επιταχύνουμε περισσότερο τη βελτίωση της διακυβέρνησης αντί να θέλουμε να αναλαμβάνουμε υπερβολικά πολλές ευθύνες ε, στην ίδια περιφέρεια, στην ίδια περιοχή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κ. Νιούτον Ντάν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση από το ελεγκτικό συνέδριο. Διαρωτώ με πώς γίνεται αυτή, αυτός ο έλεγχος. Ίσως ε, πάτε σε, κάποια από κάθε μια από αυτές τις χώρες και τα μελετάτε όλα επί τόπου. Δεν παίρνει υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν είναι πολύ δαπανηρό αυτό. Πώς το κάνετε αυτό από πλευράς ελέγχων. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να θέσω την ερώτηση. Νομίζω ότι η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ανησυχητική. Μας λέτε ότι σε 23 προγράμματα, από τα 23 προγράμματα σε διάφορες χώρες, και κάποια από τα προγράμματα αυτά έχουν προχωρήσει ιδιαίτερα όπως η Τανσανία, δεν βρήκατε παρά μόνο τέσσερα από τα 23 τα οποία είναι πραγματικά υποστηρίξιμα ενώ έχουμε δαπανίσει, αν δεν κάνω λάθος, συνολικά δύο δις και εκατοντάδες ε, ε, εκατομμύρια επιπλέον για αυτές τις μονάδες επεξεργασίας των λιμάτων. Ε, λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Έχουμε πολύ ανησυχητικά στοιχεία. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν πώς έγινε, πώς συνέβη να έχουμε 18 προγράμματα τα οποία να είναι τόσο ελαττωματικά. Πώς και δεν είδαμε λίγο νωρίτερα ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, προβλήματα στα οποία δεν υπήρξε καμία διόρθωση. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Θα κάνω κάποια αρχικά σχόλια και μετά θα είμαι στη διάθεσή σας για να δώσω απαντήσεις. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει ότι το συνέδριο ε, ε, συμφωνεί στο ότι έχουμε κάνει προσπάθειες για να πετύχουμε τους συμπεφωνημένους στόχους και ότι τα προγράμματα αυτά έχουν βελτιώσει την πρόσβαση ε, στο καθαρό νερό και τα προγράμματα έχουν προχωρήσει και βρίσκονται σε λειτουργική φάση. Τώρα για τα συγκεκριμένα ευρήματα του ελεγκτικού συνεδρίου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι στα περισσότερα προγράμματα εντοπίστηκαν σωστά οι ανάγκες και κάποιες από τις ανάγκες αυτές καλύφθηκαν. Ορισμένα προγράμματα ήταν πάρα πολύ ε, φιλόδοξα και κάποιες δευτερεύουσες ανάγκες ε, δεν μπόρεσα, ή δεν μπόρεσε η Επιτροπή να τις καλύψει. Το συνέδριο σημειώνει ότι η πλειοψηφία των προγραμμάτων δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει μέσω πρόθεσμα εκτός ε, και αν διασφαλιστεί η χρηματοδότηση εκτός ένωσης των προγραμμάτων αυτών. Εμείς θα κάνουμε εδώ την εξής παρατήρηση σχετικά με την εξωτερική λειτουργικότητα εμείς υποστηρίζουμε τις διαδικασίες κατάρτισης έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να διαχειρίζονται τις εγκαταστάσεις τους με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα. Για να διασφαλίσουμε την μελλοντική τους αηφορία και λειτουργία προσπαθούμε σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο προγραμμάτων πλαισίων στηρίζουμε κάποια προγράμματα μέσω των οποίων οι συγκεντρωτικές δομές θα μπορέσουν να διαχειριστούν τα προγράμματα αυτά στο μέλλον καθορίζοντας με σωστή αηφόρο θα έλεγα πρακτική τους τομείς αυτούς θα πρέπει να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στα εξωτερικά κόστη, στην τιμολόγηση και στους φόρους. Η τιμολόγηση από μόνη της δεν μπορεί να καλύψει το κόστος λειτουργίας. Αυτό αφορά και τις χώρες της Ευρώπης και τις χώρες της υποσαχαρικής Αφρικής, όπου υπάρχουν πολύ ε, περιορισμένες δυνατότητες σε ορισμένες από τις ε, ε, χώρες αυτές και σε ορισμένα τμήματα ευάλωτα του πληθυσμού. Προσπαθούμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε τομιακής, τομεακής φύσης διάλογο με τις χώρες αυτές ανάλογα με τις ανάγκες Λέγει το ελεγκτικό συνέδριο ότι δεν έχει δοθεί πάρα πολύ βάρος στο θέμα της επεξεργασίας των λιμάτων και της υγιεινής. Και αυτό έχει μειώσει ακόμα περισσότερο το βάρος των δραστηριοτήτων αυτών. Εδώ θα συμφωνήσουμε με το ελεγκτικό συνέδριο. Δυστυχώς συνολικά δεν έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες εξυγίανσης στο παρελθόν των υδάτων και γι' αυτό τα λαμβάνουμε υπόψη μας ε, όταν σχεδιάζουμε νέα προγράμματα ιδιαίτερα σε ημιαστικές ε, ή περιοχές της υπαίθρου. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης ότι παρά τις συνολικά ικανοποιητικές μορφές διαχείρισης η Επιτροπή δεν κατάφερε να προωθήσει την αηφορία και τη λειτουργικότητα των αποτελεσμάτων και αυτό θα πρέπει να γίνει καλύτερα μέσω των δυνατοτήτων αξιολόγησης που υπάρχουν. Εμείς απαντάμε ότι τα περισσότερα προγράμματα έγιναν δεκτά πριν από τις ομάδες ποιοτική στήριξη που δημιουργήθηκαν μετά το 2007 που επιτρέπουν την καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο των προγραμμάτων μας. Οι συστάσεις τώρα που κάνει το συνέδριο, εμείς συμφωνούμε με τις συστάσεις αυτές. Ήδη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για τη βελτίωση των διαδικασιών αυτών και θα λάβουμε υπόψη μας αυτά που λέει το συνέδριο για να προωθήσουμε στον τομέα της επιτυχίας των προγραμμάτων μας. Ευχαριστώ για τα σχόλια τα οποία κάνατε. και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένες από τις ερωτήσεις τις οποίες έθεσαν οι συνάδελφοί σας. Σχετικά με τη διατροφή. Στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να εντοπίσει προγράμματα στη διασταύρωση της διασφάλισης από τη μία υδάτινων πόρων, καθαρού νερού και από την άλλη επαρκούς ποσότητας ε, τροφίμων. Έχουμε την πρόθεση να προχωρήσουμε στην ολοκληρωμένη μορφή διαχείρισης των υδάτινων πόρων, εκεί όπου η γεωργία απορροφά τα μεγαλύτερα, τη μεγαλύτερη ποσότητα υδάτων. Τώρα, για τη δημοσιονομική στήριξη. Δεν αξιολογήθηκε. Το προσωπικό μου σχόλιο εδώ είναι ότι ε, ενημερωτικά το λέω υπάρχουν λίγες χώρες στις οποίες εμείς εργαζόμεθα επί τη βάση της στήριξης του προϋπολογισμού ε, στην υποσαχαρική Αφρική. Το χρησιμοποιούμε το σύστημα αυτό σε άλλες γειτονικέ περιοχές. Υπάρχουν κάποιες χώρες όπου εφαρμόζεται η δημοσιονομική στήριξη, όπως σαν παράδειγμα στην Μπουρκίνα Φάσο. Έχουν υπάρξει κάποιες θετικές αξιολογήσεις αυτής της προσπάθειας από το ελεγκτικό συνέδριο. Σχετικά τώρα με τη διακυβέρνηση αυτών των προγραμμάτων, τη διαχείρισή τους και το θέμα της μη χρηματοδότησης αμυγός τεχνικών προγραμμάτων. Η άποψη εδώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέγει ότι θα πρέπει να παραμείνουμε και στους δύο τομείς. Απ' τη μία να βελτιώσουμε τη διαχείριση. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι έτσι ώστε να υπάρξει συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα και επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα απαιτείται ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον και προσπαθούμε να το προωθήσουμε. Ταυτόχρονα όμως απαιτείται να παράσχουμε καθαρό νερό και να προστατεύσουμε την υγιεινή του πληθυσμού μέσω της πρόσβασης στο καθαρό νερό και της εξυγίανσης των λιμάτων. Και αυτό απαιτεί την δημιουργία και στήριξη τεχνικών προγραμμάτων. Αν κατάλαβα καλά, υπήρξε επίσης και μία ερώτηση για το πώς εμείς προχωρούμε σε κάθε μία από αυτές τις χώρες, πώς εντοπίζουμε τα προγράμματα. Ο κύριος Ντίβα έχει στήσει το λόγο. Αυτή η απάντηση πρέπει να καταχωρηθεί ως κλασικά ο τρόπος να μην απαντάτε μια ερώτηση, διότι μια δήλωση πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ας το πω έτσι φιλοδοξιών, ευχολόγια, δεν θέλουμε δηλώσεις επί πολιτικών, θέλουμε να ξέρουμε τι θα κάνετε χειροπιαστά, να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που ήδη τέθηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο. Είπατε στην απάντησή σας ότι το 2005 ξεκίνησε αυτή η διαργασία τώρα έχει λειτουργήσει και τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Τι κάνατε και τι λειτουργήσε πρακτικά χειρόπιαστα. Αυτό να μας πείτε. Όχι ευχολόγια και καταλόγους ευχών. Πρακτικά χειρόπιαστα. Υπό όρους καθημερινής ζωής ε, για να κατανοήσουμε ότι το ένα ή το άλλο βελτίωσε την κατάσταση. Τι ακριβώς έγινε α, β, γ, δ, 1, 2, 3, 4, αυτό κάναμε, τούτο, τ' άλλο, το παράλλο. Για να καταλάβουμε περί τι πρόκειται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς έχει τον λόγο, παρακαλώ. Euh, ναι κυρία Πρόεδρε πρέπει να σας ομολογήσω ότι μετά από αυτή την πρώτη σειρά απαντήσεων οι ερωτήσεις μου πολλαπλασιάστηκαν. Ε, εγώ θα ήθελα να καταλάβω τι διαδικασία ακολουθείτε. Ε, Καταρχά, όταν ξεκινάτε ένα έργο, ορίζετε τι προδιαγραφέ και στι προδιαγραφέ λέτε ότι θα προσφέρουμε ας πούμε, πρόσβαση στο νερό στην Ουαγκαντουγκού, για παράδειγμα, σε μια συγκεκριμένη συνοικία. Θα φροντίσουμε να υπάρχει πρόσβαση σε τρέχομενο νερό. Για να είναι βιώσιμο τώρα το έργο, μπορούμε να ακολουθήσουμε διάφορε μεθόδου. Αν περιλαμβάνει του πάντε, που μου φαίνεται ελάχιστη απέτηση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται τους ε, πιθανούς χρήστες που έχουν χρήματα να το πληρώσουν και αυτούς που δεν έχουν. Αν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας αυτό πρέπει να επιληθεί. Αλλά δεν θα δώσει αυτά τα χρήματα η Κομισιόν, δεν θα τα δίνει αυτά τα χρήματα επάπειρον, δεν είναι αυτή η δουλειά της Κομισιόν. Οι δικαιούχοι της αρρωγής, οι εταίροι μας δηλαδή, θα πρέπει να φροντίσουν να είναι βιώσιμα τα προγράμματα. Ε, αν το πρόβλημα είναι φορολογίας αυτό θα πρέπει να ε, αποτελέσει μέρημνα της, ε, του Δήμου της Ουαγκαντουγκού για παράδειγμα στο παράδειγμα που σας αναφέρω αλλιώς μπορεί να έχετε πολύ ωραία προγράμματα βιώσιμα ε, αν έχετε επίσης προγράμματα μόνο για αυτούς που μπορούν να πληρώσουν το νερό για να γεμίζουν τις πισίνες τους σε μια πλούσια συνοικία το ερώτημά μου είναι κατά πόσο υπάρχουν στάνταρ προδιαγραφές για όλα τα προγράμματα από την Κομισιόν. Αν σε όλα τα προγράμματα προβλέπεται πρόσβαση στο νερό για τους άπορους ως απόλυτη προτεραιότητα. Εάν τα κριτήρια, οι προδιαγραφές είναι στάνταρ, τότε μπορούν να εφαρμοστούν τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης στα διάφορα προγράμματα. Αλλιώς θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε την αξιολόγηση Κατά τη διάρκεια αυτή τη συζήτηση, ουσιαστικά, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποιε διαφορέ μεταξύ μα εδώ. Ε, καθώς συζητάμε το ζήτημα ουσιαστικά αποδεχόμαστε ότι η ανάπτυξη γίνεται από τον φορολογούμενο. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε αυτή την προσέγγιση. Το κακό εντό εισαγωγικών που έχει γίνει. Μπορεί να διορθωθεί. Αν το πρόβλημα είναι θέμα χρηματοδότησης, ε, θα πρέπει να συζητήσουμε με τον εταίρο και όταν το ελεκτικό συνέδριο και αν εδώ τώρα απευθύνονται κύριο στο ελεκτικό συνέδριο, βέβαια και στην Κομισιόν, μπορείτε να μας ορίσετε κάπως ε, πώς εκτιμάτε τη βιωσιμότητα χρονικά συγχρονικό άξονα. Να σας πω πώς την βλέπω εγώ. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα έργο το οποίο υλοποιείται το 2013. Ορίζω τις προδιαγραφές, υλοποιείται το έργο το 2016. Ξεκινάει η υλοποίησή του δηλαδή. Η φάση υλοποίηση διαρκεί ας πούμε 4 χρόνια, δηλαδή το 2020 είναι το έτος όπου έχει κλείσει το πρόγραμμα, το παραδίδουμε στον δικαιούχο της αρρωγής. Εκείνη τη στιγμή οικειοποιείται επίσημα το πρόγραμμα. Όταν τώρα κάνετε μια κριτική της βιωσιμότητας, την κάνετε το, για το 2020, το 2022, το 2025, εγώ πιστεύω ότι για να είναι πραγματικά βιώσιμο το έργο πρέπει να εξετάσετε τι γίνεται το 2030, αν βγαίνει νερό από τη βρύση το 2030. Ε, πρέπει να μας πείτε λοιπόν πώς ορίζεται αυτή τη βιωσιμότητα τι κριτήρια χρησιμοποιείται για τη μέτρησή της χρονικά. Πιστεύω είναι σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να ρίξουμε φως στις ε, κρυφές αυτές πτυχές. Merci. Ευχαριστώ. Ξαναδίνω το λόγο στην Κομισιόν ώστε να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Alors, je pas son nom. Oui, je pas son nom. Donc, monsieur. Voilà. Je m'appelle Dalamangas et je viens de DEVCO. Ονομάζομαι Δαλαμάνια και προχωρώ από την ΤΕΒΚΟ. Έχω την εντύπωση ότι η ερώτηση προοριζόταν για το ελληνικό συνέδριο, αν κατάλαβα καλά. Πρόεδρος, όχι, είναι πρώτα για εσάς, για την Κομισιόν. Για όλους, λέει ο κύριος Γκέρενς. Ε. Έχουμε ερωτήσεις για όλους σας. Τα κριτήρια αξιολόγησης, ε, φυσικά όσοι κάνουν τις αξιολογήσεις πρέπει να μας τα ε, πούν, αλλά για τις προδιαγραφές είναι η Κομισιόν και αυτοί που εκτελούν τις αξιολογήσεις πρέπει να μας μιλήσουν για τις προδιαγραφές γιατί βάσει αυτών των προδιαγραφών θα κρίνουμε ένα έργο. Η πρώτη ερώτηση είναι το τι κάναμε συγκεκριμένα για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι από το 2005 έχουμε τις ομάδες στήριξης ποιότητας. Εκεί συζητιούνται όλα τα προγράμματα και όλοι οι εμπλεκόμενοι με τα προγράμματα πρέπει να κάνουν προτάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των προγραμμάτων. Η βελτίωση των προγραμμάτων συμπεριλαμβάνει και τη βελτίωση των στόχων των προγραμμάτων, Είπα ότι πριν από το 2005 η ομάδα αυτή δεν υπήρχε. Υπήρχε λοιπόν κάποιος κάπου ο οποίος έκανε μία πρόταση και η πρόταση στην ουσία ελεγχόταν από αυτόν. Ενώ τώρα γίνεται μία ευρυτάτη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικό, σε επίπεδο ε, μηχανικό, σε επίπεδο οικονομικό. Συζητάμε το θέμα της αηφορίας των προγραμμάτων και για μένα αυτό είναι μια σημαντική βελτίωση. Υπάρχει επίσης και η διαδικασία παρακολούθησης η οποία ασκείται από τις αντιπροσωπείες μας και στο τέλος έχουμε τις αξιολογήσεις. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα το οποίο παρακολουθεί την εξέλιξη των προγραμμάτων αυτών από την αρχή μέχρι το τέλος. Αν με ρωτήσετε το τι κάναμε τον τελευταίο χρόνο ή τα τελευταία δύο χρόνια, να πω ότι τα συστήματα αυτά θα δείξουν τα ωφέλη από τη χρήση τους ε, σε λίγα χρόνια, όχι αμέσως. Δίνω τον λόγο τώρα στον κύριο Μπόστοκ του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να απαντήσω στις ερωτήσεις ξεκινώντας με τις πιο απλές. Πώς έχει προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή το συνέδριο. Κοιτάξτε, εγώ ανέλαβα το θέμα αυτό μετά από την ολοκλήρωση ενός μεγάλου ποσοστού της δουλειάς. Δέκα άτομα από το προσωπικό του ελεγκτικού συνεδρίου χρησιμοποιήθηκαν για το θέμα αυτό. Χρησιμοποιήσαμε ε, τον χρόνο εργασίας 178 ημερών ανά Εξετάσαμε αντίστοιχες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επισκεφθήκαν ορισμένα από τα προγράμματα για να δουν αυτά που θα έβλεπαν και να τα συγκρίνουν με αυτά τα οποία ε, αναγράφονται στα προγράμματα. Έτσι συνήθως γίνεται. Ποιοι ήταν οι τοπικοί εταίροι. Κοιτάξτε κύριε Γκέρενς, τοπικοί εταίροι είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα το, της παροχής καθαρού νερού, όπως επίσης και επεξεργασίας των λιμάτων. Τώρα έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της χρηματοδότησης χρηματοδοτήθηκαν άμεσα τα προγράμματα και δεν μπορούμε να σας δώσουμε περισσότερες απαντήσεις για άλλου τύπου χρηματοδοτήσεις άμεσα στον προϋπολογισμό. Τώρα για το πώς ε, και πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σταματήσει να είναι υπεύθυνη για την ε, λειτουργία των προγραμμάτων αυτών και πότε θα μεταφερθεί στους τοπικούς αν θέλετε εμπλεκομένους. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι έχει μία ευθύνη να βελτιστοποιήσει τις δυνατότητες έτσι ώστε μακροπρόθεσμα να είναι σε θέση οι τοπικοί εταίροι να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα αυτά και τα χρήματα των φορολογουμένων να είναι ωφέλιμα για μία μακρά περίοδο και όχι σύντομη περίοδο. Τώρα για την περίοδο αναφοράς ζήτησε ο κύριος Γκέρεντς να μάθει Έχουμε την ίδια περίοδο αναφοράς ε, με το Λονδίνο και το Λουξεμβούργο. Ε, όχι βέβαια. Αυτό το οποίο μπορούμε να σας πούμε είναι ότι εμείς κάναμε έναν έλεγχο το 2011, εξετάσαμε κάποια προγράμματα τα οποία είχαν ξεκινήσει στο δεύτερο ήμιση του 2000, της δεκαετίας του 2000 και είδαμε ότι κάποια από τα προγράμματα αυτά δεν πήγαιναν καλά και δεν υπήρχε και μελλοντική δυνατότητα χρηματοδότησής τους. Οπότε τώρα αν η περίοδος αναφοράς είναι 20 ή 30 χρόνια είναι λίγο αισιόδοξη και μακράν της πραγματικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε επίσης και στις ε, ομάδες ε, ποιοτική στήριξης. Ε, πράγματι, εν μέρη έχει δίκιο, συνήθως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα προγράμματα αυτά δεν υπήρχαν όταν ξεκίνησαν οι πρωτοβουλίες αυτές, αλλά πράγματι δεν είναι εντελώς σωστή εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αυτές οι ομάδες δεν ισχύουν και δεν εφαρμόζονται στον τομέα των, της επεξεργασίας των υδάτων και του μέσου για το νερό και αυτό είναι κάτι το οποίο θα αφορά πάνω από τα μισά προγράμματα που έχουμε τώρα μπροστά μας συμπερασματικά να πω ότι κάποια από τα μέλη εξέφρασαν μια κάποια λύπη για τα αποτελέσματα του ελέγχου μας. Ο εισηγητής είπε ότι μου προκάλεσε λύπη. Αλλά κοιτάξτε, εμείς σας λέμε την αλήθεια και να σας μεταφέρουμε αυτά που βρίσκουμε. Και αυτό καθιστά τις εκθέσεις μας μερικές φορές διόλου ευχάριστες. Κύριος Γκέρεντς έχει το λόγο πάλι. Έχετε δίκιο να λέτε ότι είναι η αγνάγνωση ε, ιδιαίτερα λυπηρή όταν ε, δακτυλοδεικτείται συγκεκριμένα λάθη. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να αφαιρέσουμε από την προσπάθεια αξιολόγησης κάποιες ακραίες περιπτώσεις όπου κάποιος κλέβει τα χρήματα του προγράμματος. Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό και απαράδεκτο που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να φανεί προς το κοινό ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι όλα τα προγράμματα και όλα τα λάθη που έχουν γίνει έγιναν καλή την πίστη. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κοιτάξτε, η αξιολόγηση είναι κάτι το πάρα πολύ ευαίσθητο και τίθεται εδώ το θέμα προς το ελεγκτικό συνέδριο αν έπρεπε να εφαρμόσετε τα ίδια standards στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου όλα τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα από το 2015 και μετά να έχουν μεταφέρει, μεταφέρει την οδηγία για τα ύδατα στην εθνική τους νομοθεσία. Αναρωτιέμαι αν σε αυτή την περίπτωση δεν θα αντιμετωπίζατε τις ίδιες εκπλήξεις που αντιμετωπίσατε στην υποσαχαρική Αφρική. Γιατί υπάρχουν πολλές χώρες όπου η οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν εφαρμόζεται και μιλάω για ευρωπαϊκές χώρες. Σαν παράδειγμα ε, η διασφάλιση της ε, τιμολόγησης ε, έτσι ώστε ο καταναλωτής να καταστήσει το πρόγραμμα αυτό βιώσιμο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε κάπως σχετικιστές εδώ. Γιατί αν δεν εμφαρίνουμε ε, μια μεγαλύτερη γνώση των προβλημάτων και να, αν δεν κάνουμε προτάσεις για να βγούμε από τα προβλήματα αυτά, τότε δεν θα είμαστε αξιόπιστοι. Εγώ ίδιος έχω δει από κοντά τέτοιου είδους αξιολογήσεις ε, και η πρακτική στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν να προστίθενται ορισμένα προγράμματα διαχείρισης στα προγράμματα τα οποία δεν είχαν ικανοποιητική εξέλιξη. Αυτό γίνεται στον τομέα των νοσοκομείων και στον τομέα της πρόσβασης στο καθαρό νερό. Στα νοσοκομεία, σαν παράδειγμα, χρειάστηκε να γίνουν αξιολογήσεις ε, για τη λειτουργία νοσοκομιακών μονάδων που δεν υπήρχε επαρκή χρηματοδότηση. Μπορείτε να μου πείτε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όπου τα νοσοκομεία να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ακόμα και στις χώρες ε, της υποανάπτυξη πρέπει να επιδοτούμε τέτοιου προγράμματα και αυτό θέτει σε αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα και την αηφορία των προγραμμάτων. Αυτό δεν είναι σωστό. Θα πρέπει μήπως ε, να σκεφτείτε κι εσείς αν δεν είναι ιδιαίτερα σκληροί η αξιολόγηση την οποία κάνετε και μήπως υπάρχουν κάποιες εξηγήσει για την κατάσταση αυτή. Το θέμα είναι βέβαια πώς θα διορθώσουμε τα πράγματα. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες μπορεί να αναλυφθούν τους επόμενους μήνες έτσι ώστε τα προγράμματα τα οποία έγιναν αντικείμενο κριτικής να μπορέσουν να διασωθούν. Και τα προγράμματα αυτά μπορεί να ενταχθούν σε μια τροχιά θα έλεγα αποδεκτή. Αυτό είναι το θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ θέτουμε πολύ σημαντικά ερωτήματα όσον αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του πολιτικών ελέγχων, τη συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα ξαναδώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να απαντήσει στις τελευταίες παρατηρήσεις του κ. Γκέρενς και ενδεχομένως για τη δική μας ε, Επιτροπή ε, θα μπορούσε να επινοηθεί κάποια αντόκ διαδικασία ελέγχου σε αυτήν την πολύ ανησυχητική κατάσταση. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Κομισιόν πριν ολοκληρώσει τη γνωμοδότηση της η κυρία Ζαβόσκα. Ε, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, όσον αφορά την παρατηρήση του ελεγκτικού συνεδρίου για τα προγράμματα διευκόλυνσης για τα, για τα ύδατα που δεν περνάει από την ομάδα υποστήριξης ποιότητας. Αυτά τα προγράμματα έγιναν αποδεκτά μέσω μιας πιο σκληρής διαδικασίας μέσω της κλήσης για υποβολή προσφορών. Αξιολογήθηκαν από πολλούς. Δεν είναι προγράμματα τα οποία διαμορφώθηκαν από την Κομισιόν. Είναι προγράμματα ο ομικρών ή τοπικών ε, κυβερνήσεων που προτάθηκαν, αξιολογήθηκαν κτλ. Αυτό για να μην δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση. Τώρα όσον αφορά το ζήτημα των προγραμμάτων που δεν επιτυχάνουν τους στόχους τους. Θα ήθελα να σας πω για παράδειγμα, ένα παράδειγμα που μου έρχεται στο νου, ένα πρόγραμμα στην Τανζανία, όπου στόχος ήταν η οικοδόμηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων. Δεν κατασκευάστηκε, συνεπώς δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι. Δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι όμως γιατί ο προϋπολογισμός δεν ήταν επαρκής. Οικοδομήσαμε λοιπόν αυτό στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας με μια δεύτερη φάση. Το πρόγραμμα της πρώτης φάσης δεν ήταν επιτυχές. Αλλά το θέμα ήταν εδώ, θέμα χρηματοδότησης που εντοπίσαμε αργότερα, στη μεταγενέστερη φάση. Ε, αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο μας λέει ότι τα πράγματα δεν είναι άσπρα ή μαύρα. Πρέπει να εξετάζουμε κατά περίπτωση τι έγινε καλά, τι δεν έγινε καλά, τι πέρασε καλά, τι όχι, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να καταλήξουμε σε ένα πιο ικανοποιητικό επίπεδο. Δεν είναι εύκολο όμως να λέμε αυτή τη στιγμή ότι το 80% των προγραμμάτων ήταν ε, καταστροφικά, ότι τα δε ποσοστό δεν πέτυχε τους στόχους. Είναι πολύ πιο σύνθετη η κατάσταση. Είναι πολύ πιο περίπλοκο να περιγράψει κανείς ε, τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης. Ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Ζάμποσκα για να κλείσει και να μας κάνει προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους θέλω να τους ευχαριστήσω που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση ήταν πραγματικά διεξοδική, περιεκτική και μεγάλης αξίας. Χαίρομαι λοιπόν για το γεγονός ότι η εντύπωση των συναδέλφων σε σχέση με την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ε, και ε, τα όσα μπορέσαμε να αποκομίσουμε ήταν ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Η διασφάλιση των πτυχών της υγείας είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Ένα ιδιαίτερα δυσχερές πρόβλημα είναι περίπλοκη και σύνθετη η απάντηση ως λύση που πρέπει να δοθεί και πρόκειται για ένα τομέα όπου θα πρέπει να βοηθήσουμε και να συνεισφέρουμε και όσο πιο περίπλοκο είναι το θέμα και σε σχέση με μια περιφέρεια ή περιοχή, τόσο πιο δύσκολη είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο κύριος Γκέρενς αναφέρθηκε σε, στο θέμα δικτών, πως δίκτες θα μπορούσαν να βοηθήσουν για την αξιολόγηση αυτού του προβλήματος. Θα πρέπει όμως να μπορέσουμε να το συζητήσουμε σε μια άλλη χρονική στιγμή και να δούμε κριτήρια αναφοράς, στοιχεία αναφοράς για τη διαθεσιμότητα αυτών των ε, δράσεων. Και τα κονδύλια τα οποία σε 10 χρόνια για παράδειγμα ε, από το 2001 μέχρι το 2010 και θέλω να το τονίσω αυτό σε αυτή την περίοδο κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύθηκαν για την ε, τον καθαρισμό του νερού σε ένα συνόλου ενός δις, ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Είναι ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό. Αν δούμε τώρα τα κριτήρια για τη διαθεσιμότητα και την ε, παραγωγή του καθαρού νερού, πόσιμου νερού, θα ήθελα να αναφέρω και κάποια θέματα που αφορούν προσωπική πείρα. Τα κριτήρια για τα, τη διάθεση κονδυλίων, για την ε, διάθεση αντλειών ή για τη δημιουργία πηγαδιών προς άντληση νερού ήταν τα εξής. Προβλεπόταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα είχαμε πενταετή πείρα και πρακτική ε, εμπειρία σε σχέση με τη διαθεσιμότητα, την δυνατότητα ενός παρόχου για τη δημιουργία μιας τέτοιας ε, μονάδας. Κάνουμε λόγο εδώ για τις πιο φτωχές περιοχές και τις πιο φτωχές χώρες. Είναι αδύνατο να βρεθούν άτομα που να έχουν τέτοιου είδους πείρα, που να ξεπερνούν και μια πενταετή περίοδο όσον αφορά την ε, δημιουργία, την διάθεση τέτοιου είδους αντλειών και τέτοιου τέτοιου είδους πηγαδιών. Πρέπει λοιπόν πιο συνεκτικά και με μεγαλύτερη συνέπεια να μπορούμε να εργαζόμαστε. Και αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους από την άλλη πλευρά, τους συναδέλφους που συμμετείχαν. Και είμαι φυσικά στη διάθεσή σας αν έχετε άλλες παρατηρήσεις ή ερωτήσεις για τη γνωμοδότησή μου. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ζάμποσκά, Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών για τη γνωμοδότηση της κυρία Ζαμπορσκά είναι η 31η Ιανουαρίου στι 3 η ώρα μετά μεσημβρίας και ότι θα ψηφίσουμε αυτή τη γνωμοδότηση στις 19 Φεβρουαρίου. Τώρα θα περάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια θα επανέλθουμε στην έκθεση του κ. Κάσμαν Περνάμε στο σημείο 9, το οποίο εξετάζουμε αργότερα λόγω της καθυστέρησης ε, των σιδηροδρόμων. Θα εξετάσουμε τώρα τη Συμφωνία Αντιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαδαγασκάρης. Και δίνω χωρίς καλή καθυστέρηση το λόγο στον εμπειρογνώμονά μας που συνέταξε αυτή τη γνωμοδότηση την κυρία Ιζαμπέλα Λέβεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μόλις ήρθε από την Επιτροπή Αλίας και πολλοί είχαν προβλήματα με τα τρένα και τις πτήσεις, με όλες τις χιονοπτώσεις όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, η γνωμοδότησή μου για τη Συμφωνία Αλληλευτικής σύμπραξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαδαγασκάρης αφορά ένα νέο πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαδαγασκάρης. Αυτό το πρωτόκολλο καλύπτει μια διετή περίοδο που ξεκινάει 31 Ιανουαρίου 2013. Εγώ ήμουν εισηγήτρια της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας για τη μελλοντική εξωτερική διάσταση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής που ψηφίστηκε το περασμένο φθινόπωρο στην Ολομέλεια και εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Ένα από τα κυριότερα σημεία είναι ότι χρειαζόμαστε συνοχή πολιτικής όσον αφορά την ανάπτυξη μεταξύ της αλληλευτικής πολιτικής και των αναπτυξιακών πολιτικών. Όπως γνωρίζετε, οι συμφωνίες αλληλευτικής σύμπραξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποτελέσει το αντικείμενο κριτικής μέσα στα τελευταία χρόνια αναφέρεται ότι εκμεταλλευόμαστε τους πόρους των ε, τρίτων χωρών και ότι δεν σεβόμαστε κάποιες θεμελιώδεις αρχές ε, βιωσιμότητας ε, χρήσης διακυβέρνησης και ακόμη και δημοκρατίας, ότι ουσιαστικά κάνουμε δουλειές με χώρες που παραβιάζουν τις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας για την εκθέση μου ήταν πολύ καλό και στο εξή ελπίζω ότι όλες οι συμφωνίες ελευτικής σύμπραξης θα ακολουθούν αυτές τις ε, πολύ ικανοποιητικέ αρχές. Θα επανέλθω σε αυτό. Για να μιλήσουμε τώρα για αυτό το συγκεκριμένο πρωτόκολλο με τη Μαδαγασκάρη, είναι μια τυπική συμφωνία για τον τόνο. Συνήθως αυτές οι συμφωνίες δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα της μικρή, μικρής κλίμακα, τη μικρής κλίμακας αλληλεία σε αυτές τις χώρες διότι ο τόνος αλλοιεύεται σε μεγάλες αποστάσεις από την ακτή. Ο τόνος επίσης ε, μεταναστεύει σε μεγάλο βαθμό. Ουσιαστικά τα σκάφη πρέπει να ακολουθούν το είδος αυτό σε μεγάλες περιοχές. Αυτό το πρωτοκόλλο λοιπόν με την Μαδαγασκάρη είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον Ινδικό ωκεανό. Αυτό το νέο πρωτόκολλο αυξάνει το τμήμα που προορίζεται για το τομεακή στήριξη από 132.000 ευρώ ετησίως σε 550.000 ευρώ το χρόνο και ο τομεακή στήριξη όπως γνωρίζετε προορίζεται για την ε, αυξήσει της παρακολούθησης του ελέγχου, της επιτήρησης και της επιστημονικής αξιολόγησης και ούτω, και καθεξής και για την υλοποίηση της διαχείρισης ε, των ε, τόπων αλληλείας και πιστεύω ότι αυτή η αύξηση συγκεκριμένη συμφωνία είναι καλοδεχούμενη διότι οι εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι υπάρχει ελάχιστη επιστημονική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαδαγασκάρης και υπάρχει τεράστιο περιθώριο βελτίωσης. Και η Μαδαγασκάρη χρειάζεται επίσης να βελτιώσει το επιστημονικό της έργο ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες συλλογή δεδομένων της Επιτροπής Ινδικού Ωκεανού. Ένα ανησυχητικό κομμάτι αυτού του νέου πρωτοκόλου είναι η νέα ρήτρα εμπιστευτικότητας. Πρόκειται για κάτι νέο στα πρωτόκολλα των Συμφωνιών Αλληλευτικής Σύμπραξης. Το έχω δει αυτό το στοιχείο ήδη μερικέ φορέ και θα ήθελα να το αναφέρω ξανά ενώπιον αυτή τη Επιτροπής. Είναι ανησυχητικό όταν έχουμε μιλήσει τόσο πολύ για διαφάνεια και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και ότι όλοι πρέπει να μπορούν να βρουν ε, τα περισσότερα δυνατά στοιχεία για την αλληλεία στα υδατά τους και εμείς εισάγουμε αυτή τη νέα ρήτρα εμπιστευτικότητας που λέει ότι ανα πάσα στιγμή όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αλληλευτικές τους δραστηριότητες στα ύδατα της Μαδαγασκάρης θα θεωρούνται εμπιστευτικά. Ανα πάσα στιγμή όλα τα στοιχεία. Καλύπτει δηλαδή τα πάντα. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να το επικρίνουμε και να αλλάξει στα πρωτόκολλα αυτά. Αυτό που καλωσορίζουμε είναι τη ρήτρα αποκλειστικότητα, έτσι ονομάζεται. Αυτό σημαίνει ότι όταν υπάρχει μια συμφωνία αλληλευτική σύμπραξη σε μια τρίτη χώρα, όλα τα σκάφη τη Ευρώπη που έχουν το δικαίωμα αλληλεία πρέπει να ε, εντάσσονται στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Δεν γίνονται δηλαδή ιδιωτικέ συμφωνίες μεταξύ ιδιωτών. Επίσης υπάρχουν και νέες διατάξεις όσον αφορά την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων που καλωσορίζουμε ιδιαίτερα. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ως πολύ καλό στοιχείο είναι αυτή η συμπεριλήψη των ορίων αλληλεία καρχαριών. Δεν τους μετρούσαμε τους καρχαρίες στο παρελθόν. Αν κοιτάξετε λοιπόν τα στοιχεία αλίευσης, τα παράπλευρα αλίευματα καρχαριών ανέρχονταν έως και στο 55% των αλίευμάτων και οι καρχαρίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν κίνδυνο, τεράστιο κίνδυνο εξάλληψης και αυτό το πρωτόκολλο λοιπόν επιβάλλει περιορισμό στα αλίευματα καρχαριών και μάλιστα αναφέρεται και σε κάποια είδη καρχαριών που αποκλείονται ρητά απαγορεύεται να αλλιεύονται πέντε είδη καρχαριών. Το θεωρούμε πολύ θετικό αυτό το σημείο και θα θέλαμε αυτό να συμπεριλαμβάνεται και στα μελλοντικά πρωτόκολλα αλληλείας με άλλες χώρες. Επανέρχομαι τώρα στην εισαγωγή μου όσον αφορά τη συνοχή πολιτικής για την ανάπτυξη και τις υποχρεώσεις ε, της συνθήκης του αρθρού 208 της Συνθήκης Λισαβόνας ε, που αφορούν την συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Το 2009, λοιπόν, μετά από το πραξικόπημα στη Μαδαγασκάρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέστηλε την αναπτυξιακή συνεργασία με τη Μαδαγασκάρη. Σύμφωνα με το αρθρό 96 της Συμφωνίας του Κοτονού. Έκτοτε ε, έλαβε χώρα πολιτικός διάλογος με τη Μαδαγασκάρη, για το πώ θα μπορούσε να αποκατασταθεί η δημοκρατία και ο σεβασμός των ανθρωπινών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στη χώρα αυτή. Παρότι λοιπόν αυτό το νέο πρωτόκολλο περιλαμβάνει μία παράγραφο, ένα άρθρο, το άρθρο 8 8γ, όπου αναφέρει ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιληφθεί παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 της Συμφωνίας του Κοτονού και βάσει της διαδικασίας των άρθρων 8 και 96 τη συμφωνία σε αυτή την περίπτωση, όλες οι δραστηριότητες καφών της Ευρωπαϊκή Ένωσης στα νερά της Μαδαγασκάρης θα ανασταλούν. Θα διακοπούν. Είναι πολύ περίεργο ότι διαπραγματευόμαστε μια συμφωνία λέγοντας ότι θα τη διακόψουμε σε περίπτωση παραβιάσεων του άρθρου 9 της συμφωνίας του Κοτονού, ενώ αυτή η χώρα τελεί υπό αναστολή λόγω παραβίαση αυτού του άρθρου. Παρότι δηλαδή αυτή η πτυχή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σε αυτό το πρωτόκολλο και εγώ τη στηρίζω, δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορούσε αυτό το κοινοβούλιο να επικυρώσει αυτή τη συμφωνία, ενώ ισχύει το άρθρο 96 της συμφωνία του Κοτονού. Αυτή η Επιτροπή, θυμάμαι, πριν τα Χριστούγεννα έκανε μια συζήτηση για, τις, ε, για τη Συμφωνία Ελευτικής σύμπραξη με την Κιουίνε Μπισά, όπου εμπίπτει επίση το άρθρο 96 τη Συμφωνία του Κοτονού και τότε αποφασίσαμε η συγγήτρια κυρία Μάισνερ δεν ήθελε να συνεχίσει με τη γνωμοδότηση λόγω αυτής της συμφωνίας, λόγω της διακοπής συνεργασίας με τη Γουινέα Μπισάου. Και το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της Μαδαγασκάρης. Και τώρα η Κομισιόν ξέρω θα πει ναι, έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδο στη Μαδαγασκάρη και αναμένουμε να λάβουν χώρα εκλογές κάποια στιγμή μέσα στην Άνοιξη. Ωραία είναι όλα αυτά. Μετά τις εκλογές, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ναι σε αυτή τη συμφωνία, αλλά αυτό που προσπαθώ να πω εγώ εδώ στη γνωμοδότησή μου είναι ότι ότι θα πρέπει να προτείνουμε στην Επιτροπή Αλίας να αρνηθεί να δώσει την έγκρισή τη έω ότου έχουν λάβει χώρα δημοκρατικές εκλογές στη Μαδαγασκάρη και εφόσον είχε αποκατασταθεί η δημοκρατική τάξη. Δεν υπάρχει λοιπόν σε καμία περίπτωση κάτι το οποίο να λέγει ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε με αυτή την πρόταση ήδη από εφέτος. Υπήρξαν περιπτώσεις τις οποίες το Κοινοβούλιο δεν έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του παρά ένα χρόνο μετά από την ε, θέση σε λειτουργία των αλλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω των προκαταρτικών πρωτοκόλων, κάτι το οποίο ισχύει και σήμερα. Δεν θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν την σύμφωνη γνώμη μας αν δεν γίνουν εκλογές. Είναι βασική αρχή, πρέπει να εμείνουμε αν είχε εφαρμοστεί το 96 της συνθήκης του Κοτονού, δεν θα υπάρξει σύμφωνη γνώμη που να λέει ότι θα πρέπει να διακοπούν αυτές ε, οι αλλιευτικές δραστηριότητες αν το 9 της συνθήκης του Κοτονού δεν έχει γίνει σεβαστό και σημειούται θεμελιώδης παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λοιπόν, αυτά. Περιμένω τις απόψεις των ε, σκιωδών εισηγητών από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Υποστηρίζω τη γνώμη της κυρίας Λεβίν ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε τη συμφωνία αυτή εφόσον η Μαδαγασκάρη ε, εντάσσεται στα πλαίσια του άρθρου 96. Αυτό είναι σαφές και δεν μπορούμε επίσης να συμφωνήσουμε με τη ρήτρα απορρίτου γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος τεχνικά δεδομένα για την αλληλεία να αποκρύβονται από την κοινή γνώμη. Και γι' αυτό θα ζητήσω, όπως το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα ζητήσω τη δυνατότητα εγώ σαν πρόεδρος να έχω πρόσβαση σε όλες τις επιστημονικές πληροφορίες τις οποίες έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δίνω το λόγο στον κύριο Κάσμαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν είμαι εγώ εισηγητής των σοσιαλιστών για αυτό το θέμα, όμως πρέπει να πω ότι και ζητώ συγγνώμη για την καθυστερημένη αφήξή μου. Έχοντας ακούσει το τελευταίο τμήμα της παρουσίασης, Ω συζητή για την αναθεώρηση της Συμφωνίας ε, Κοτονού συμμερίζομαι τις ανησυχίες που εκφράζει η κυρία Λεβέα ιδιαίτερα, ιδιαίτερα κιόλα. <clears throat> σε σχέση με τον διάλογο που πρέπει να επιτευχθεί για την διακόπτη ομιλητή. ιδιαίτερα για τα, τις καταχρήσεις, τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σίγουρα από την πλευρά μας αυτό είναι αν, ανεπαρκές και αναποτελεσματικό και η ρήτρα που αναφέρεται αναφέρεται συγκεκριμένα σε θέματα αμοιβαίων ανησυχιών και μελημάτων. Και η άλλη πλευρά, αυτό το οποίο πρέπει να πει η άλλη πλευρά από πλευρά ή του ΑΚΕ, ότι αυτά τα θέματα δεν είναι θέματα τα οποία να μας απασχολούν. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει διάλογος. Απόλυτα λοιπόν καλωσορίζω και προσωπικά εγκρίνω την προσέγγιση της εισηγήτριας της κυρίας Λεβίν και προσβλέπω στο να διαμορφωθούν συζητήσεις από πλευρά σοσιαλιστών για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα για την ενίσχυση των αρχών της Συμφωνίας του Κοτονού για αυτά τα θέματα που πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικές διότι είναι ατελείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εσείς τώρα έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την εισηγήτρια κυρία Λεβίν. Η Ιζαμπέλ Λεβίν ιδιαίτερα κατέστησε σαφές γιατί εμείς ως Επιτροπή Ανάπτυξης πρέπει να μεριμνήσουμε αυτή η συμφωνία να απορρίπτεται μέχρι ότου να υπάρξουν δημοκρατικές εκλογές που θα έχουν διεξαχθεί στη Μαδαγασκάρη προηγούμενα. Θέλουμε επίσης και την διαδικασία του εκδημοκρατισμού να την υποστηρίξουμε. Όμως έναντι της Μαδαγασκάρης πρέπει να πιέσουμε, να ασκήσουμε πίεση και όταν πολιτική συνεκτικότητα και συνέπεια Θέλουμε να έχει αποτελεσματικότητα για την πολιτική για την ανάπτυξη, όπως και στην περίπτωση Γκινέα Μπισάου, όπως και τώρα στη Μαδαγασκάρη πρέπει να ασκήσουμε πίεση. Με σαφέστατο τρόπο να πούμε έναντι της Επιτροπής Αλίας ότι εμείς η Επιτροπή Ανάπτυξης παραμένουμε στα κριτήρια τα οποία θεωρούμε ότι είναι σημαντικά. Να είναι σεβαστά τα δικαιώματα του ανθρώπου, να υπάρξει εκδημοκρατισμός, το κράτος δικαίου να εγγυάται, να μπορεί να εγγυηθεί. Γι' αυτό τον λόγο απορρίπτουμε μια τέτοια συμφωνία μέχρι ότου θα έχουν διεξαχθεί προηγούμενα όμως εκλογές στη Μαδαγασκάρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα επανέλθω σε όλα όσα υπογράμμισε η κυρία Λεβεν όσον αφορά το τι είναι αποδεκτό σε αυτό το νέο πρωτόκολλο που εγώ θα ονόμαζα μεταβατικό και που έχει συσταθεί για δύο χρόνια, αλλά θα ήθελα να μπω σε κάποιες λεπτομέρειες για τα δύο σημεία που φαίνεται να παρουσιάζουν δυσκολίες για την Επιτροπή σας. Το πρώτο αφορά αυτή τη ρήτρα εμπιστευτικότητα. Πρόκειται για μια νέα ρήτρα. Δεν τη χρησιμοποιούμε για πρώτη φορά, αλλά είναι νέα. Υπάρχει ήδη σε άλλες συμφωνίες, ε, μάλιστα συμφωνία με τη Μοζαμβίκη, με το Μαυρίκιο επίσης σκοπός ύπαρξης αυτής της ε, ρήτρα είναι να μην καθιστά ασαφείς τις πληροφόριες ε, σε σχέση με την αλλιευσία από ευρωπαϊκά σκάφη. Προβλέπει απλά την προστασία των δεδομένων σεβόμενη ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις των ευρωπαϊκών ευρωπαϊκών φορέων δυνάμει των διαφορών κανονισμών που έχουν εφαρμογή. Για παράδειγμα, ο κανονισμό που σχετίζεται με το VMS, το Vessel Monitoring Scheme, το σύστημα παρακολούθηση σκαφών. Αυτή η ρήτρα, θα ήθελα να σας επισημάνω, δεν ε, έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις ε, που έχουν υλοποιηθεί από την CTOI, τον Περιφερειακό Οργανισμό Αλίας, που ρυθμίζει τα μεταναστευτικά είδη στην περιοχή. Αυτό ήθελα να υπογραμμίσω. Το δεύτερο, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η ρήτρα σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζει τις εθνικές αρχές της Μαδαγασκάρης καθώς και τις αρχές των δικών μας κρατών σημαίας των σκαφών που αλλιεύουν εκεί να λάβουν πληροφορίες όσον αφορά τη δραστηριότητα των σκαφών. Τονίζω μάλιστα ότι ορισμένα αυτά τα στοιχεία σχετίζονται απλά και μόνο με την ασφάλεια αυτών των σκαφών. Όλες λοιπόν οι πληροφορίες που επιτρέπουν να εκτιμά κανείς ακόμη και δημοσίως ε, την αλλιευτική προσπάθεια που έχει αναπτυχθεί, που, πώς και πότε, Όλες αυτές οι πληροφορίες παρέχονται, αλλά τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των σκαφών πρέπει να προστατεύονται όπως συμβαίνει ήδη και σε άλλους κανονισμούς. Δεν είμαστε κατά της διαφάνειας, αλλά μετά από κάποιο σημείο η διαφάνεια αυτή υπάρχει κίνδυνος να ζημιώσει τις ε, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Το δεύτερο που θέλω να αναφέρω το κλίμα των σχέσεών μας με τη Μαδαγασκάρη σε καμία περίπτωση οι διαπραγματευτές που είχαν αναλάβει τη διαπραγματεύση αυτής της συμφωνίας σε καμία περίπτωση δεν προσπάθησαν να παραβιάσουν αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί ή να θεωρήσουν ότι έχριζε η χώρα. ιδιαιτερη αντιμετωπιση έχει διακοπεί η αναπτυξιακή βοήθεια, όπως τόνισε η κυρία Πρόεδρος. Ήθελα να αναφέρω δύο πράγματα, ότι ουδέποτε και ποτέ, ούτε στις Βρυξέλλες, ούτε στην Ταναναρίβη, οι υπηρεσίες της Κομισιόν που έχουν επιφορτιστεί με αυτή τη διαπραγμάτευση δεν χωρίστηκαν από τους συναδέλφους του ΕΕΣ. Μεριμνούσαν ώστε να τηρούνται τα όρια που έχετε αναφέρει σε αυτή την άσκηση. Δεύτερον, έχουμε ένα, θα έλεγα, φρέσκο νέο για κάποιους. Τη δήλωση της κυρίας Άστον το περασμένο Σάββατο. Μπορώ να σας δώσω το σχετικό έγγραφο αυτή η δήλωση φαίνεται να δηλώνει ότι οι αρχές της Μαδαγασκάρης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι οι εκλογές όπως φαίνεται θα λάβουν χώρα όπως φαίνεται σε ειρηνικό περιβάλλον το Μάιο. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ κατά πόσο μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το Μάιο για να πούμε για να πει η δική σας επιτροπή ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να διακοπεί, να μην εφαρμόζεται μέχρι εκείνη τη στιγμή. Απλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στόχος αυτών των συμφωνιών ο στόχος αυτών των συμφωνιών δεν είναι ο ίδιος με το στόχο της αναπτυξιακής βοήθειας. Εδώ μιλάμε για μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός παράκτιου κράτους σημαντικού παραγοντά στον Ινδικό ωκεανό, σημαντικού κράτους στον Ινδικό ωκεανό για την βιώσιμη εκμετάλλευση δυνάμει των κανόνων που ανέφερε η κυρία Λέβεν και που αναφέρονται στην εκθεσή τη όσον αφορά την εξωτερική διάσταση με δημοκρατικό τρόπο, όπως είπε η κυρία Λέβεν, και με τρόπο ισορροπημένο. Έχουμε λοιπόν δύο επιλογές Ή καθόλου συμφωνία και σε αυτή την περίπτωση δεν στέλνουμε κανένα ευρωπαϊκό πλοίο στα ύδατα αυτά, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα για τις αρχές της Μαδαγασκάρης ότι δεν θα έχουν μέσα, διότι το υπενθύμισε η κυρία Λόβεν όσον αφορά την τομεακή στήριξη. Αυτή η συμφωνία πραγματικά προσφέρει εξαιρετικά ωφέλιμα εργαλεία για την αλληλεία στα νερά τη Μαδαγασκάρης. Δεν είμαστε μόνο εμεί αυτοί που επωφελούμαστε. Χρειάζονται και αρχέ τη Μαδαγασκάρης μέσα και οικονομικά μέσα για να μπορούσουν να εφαρμόσουν παρακολούθηση, να μπορέσουν να αποκομίσουν επιστημονικά ωφέλη για να δραστηριοποιηθούν καλύτερα. Ε, βάσει και των δραστηριοτήτων των περιφερειακών οργανισμών αλίας. Δεν έχω άλλη να πω. Καταλαβαίνω τη θέση σας, ε, κύριε Λέβεν, αλλά να προσθέσω στη ζυγαριά και αυτό το στοιχείο ότι η διακοπή, η αναστολή αυτής της ε, συμφωνίας δεν θα βοηθήσει απαραίτητα τη βιώσιμη αλία στα νερά της Μαδαγασκάρης. Κύριε Λέβιν, κύριε Κάσμαν, ζητήστε πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, σύντομο. Θα ήθελα να πω κάτι το οποίο είναι προφανέ. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια υιοθετήσαμε ένα IPA, το οποίο δεν καλύπτει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν σέβεται τις βασικές μας αρχές. Αν το αγνοήσουμε αυτό στο μέλλον, τότε τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου ε, δεν θα παίζουν κανένα ρόλο και θα τα αγνοούμε στην πρώτη φάση για να τα πετύχουμε υποτίθεται σε μια ιστερότερη φάση. Αυτά θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τις διαπραγματεύσεις μας εξ αρχής και όχι μόνο μετά την ολοκλήρωσή τους. Νομίζω ότι αυτό που το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραβιάσουμε τις αρχές μας. Κυρία Λεβίν. Ευχαριστώ κύριε Κάσμαν, είπατε ακριβώς αυτό το που ήθελα και εγώ να πω. Η Επιτροπή λέει ότι έχουμε δύο επιλογές. Ή θα έχουμε συμφωνία ή δεν θα έχουμε συμφωνία. Και θα αφήσουμε τους άλλους να αλλιεύουν στα ύδατα αυτά. Και εμείς έχουμε δύο επιλογές λοιπόν. Ή θα ακούσουμε και θα σεβαστούμε τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες έχουμε συμφωνήσει ή δεν θα το κάνουμε. it's, it's σε κάποιες περιπτώσεις το θέμα αυτό, η ερώτηση αυτή είναι, τίθεται με σοβαρό τρόπο και σε άλλες όχι, αν η συνέπεια θα είναι μόνο αποκλεισμό αποκλεισμός μας από ορισμένα αλλιεύματα κτλ. Θα πρέπει εμείς να πιέσουμε τις χώρες αυτές να αποκαταστήσουν την δημοκρατία. Αυτό είναι ένα μέσο το οποίο θα πρέπει να, αντοασκήσουμε το ασκήσουμε χωρίς εξαιρέσεις. Θα ήταν ένα κάκιστο μήνυμα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης το να, μην το να δώσουμε μάλλον τη σύμφωνη γνώμη μας χωρίς δημοκρατικές εκλογές. Το ότι υπόσχονται να κάνουν τις εκλογές το Μάιο είναι ένα καλό βήμα και ελπίζω να ακολουθήσουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρος και ο τέος πρόεδρος δεν θα είναι υποψήφοι στις εκλογές αυτές. Ένα πρώτο καλό βήμα λοιπόν. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλά και ελπίζω να έχουμε μία αηφόρο διαχείριση των μαλλιευμάτων στον Ινδικό. Δεν θα το πετύχουμε αυτό έτσι κι αλλιώς αν κάνουμε συμφωνίες με δικτατορίες και με ανεύθυνες πολιτικές ηγεσίες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν είναι ο δρόμος αυτός που θα οδηγήσει στην αηφορία στην αλληλεία. Ευχαριστώ για τις απόψεις όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ και εγώ λέει η Πρόεδρος. 28 Ιανουαρίου 12η μεσημβρινή για την κατάθεση των τροπολογιών και ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση της κυρίας Λεβίν είναι στις 19 Φεβρουαρίου. Περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα πρέπει να τελειώσουμε μέσα σε 20 λεπτά. Η αρχή υποχρέωση, αν θέλετε, του ΟΗΕ για την ευθύνη προστασίας Δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Κάσμαν, ο οποίος είναι ο εισηγητής μας για το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Κάσμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς εσάς και την Επιτροπή γιατί ήσασταν ευέλικτοι ε, στο χρονοδιάγραμμα φαίνεται ότι τα χιόνια εκπλήσουν ακόμα και τις βόρειες χώρες και γι' αυτό καθυστερούν τα το ένα μας. Ευχαριστώ εδώ την Αν Μακφάβλαν και τις υπηρεσίες πάντως για τη βοήθεια. Βλέποντας όλους αυτούς που φεύγουν από την αίθουσα, ε, καταλαβαίνω ότι δεν θα χρειαστούμε και τα 20 λεπτά. Η γνωμοδότηση αυτή, ζητώ συγγνώμη, είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα, θα είναι διαθέσιμη και σε όλες τις άλλες γλώσσες πριν περάσουμε στην επόμενη σημαντική συζήτηση. Η ευθύνη λοιπόν για την προστασία, το R2P στα αγγλικά, δημιουργήθηκε μετά από την αποτυχία της διεθνούς κοινότητας να προστατεύσει τους πληθυσμούς της Ρουάντα. Εκείνη την εποχή ο κύριος Σανάνα είχε θέσει το ερώτημα πότε θα παρέμβει η ανθρώπινη κοινότητα για την προστασία των πληθυσμών. Δυστυχώς το ερώτημα αυτό τίθεται συστηματικά από τότε σε σχέση με γεγονότα όπως στη Συρία αλλά και αλλού. Η ευθύνη για την προστασία λοιπόν είναι μια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών που καθιερώθηκε το 2005 5 συγγνώμη, θέτει ορισμένες αρχές, λέγει ότι η κυριαρχία η εθνική δεν είναι μόνο ένα δικαίωμα, αλλά είναι και μια ευθύνη και ένα καθήκον και ε, το άρθρο 4 και 5 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη και την τιμωρία ε, εγκλημάτων όπως η εθνική κάθαρση, η γενοκτονία κτλ. Ε, γενικά ε, εγκλήματα μαζικής καταστροφής. Ε, δυστυχώς και αυτά τα έχουμε γνωρίσει. Η ευθύνη λοιπόν για προστασία έχει τρεις πυλώνες εισαγωγικά. Πρώτον, το κράτος έχει την ευθύνη να προστατεύσει τους πληθυσμούς από μαζικές δολοφονίες. Η διεθνής κοινότητα έχει την υποχρέωση να βοηθήσει το κράτος αυτό να φέρει σφαίρα στην υποχρέωσή του και τέλος, το πιο δύσκολο, αν η χώρα αποτύχει ε, την προστασία αυτή και έχουν αποτύχει τα ειρηνικά μέτρα, η διεθνής κοινότητα έχει την ευθύνη μέσω ε, υποχρεωτικών αναγκαστικών μέτρων όπως οι στρατιωτικές κυρώσεις να παρέμβει με τελευταία πλέον την προσφυγή στην χρήση των όπλων. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ανέλαβε την πρωτοβουλία να καταθέσει την πρόταση αυτή, κάνοντα συστάσεις προς την Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων σε συζητήσει που θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Εγώ και οι υπηρεσίε εγώ Ρενό, πολιτικό σύμβουλο, συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της ΕΚΟ και της Υπηρεσίας Εξωτερικών Σχέσεων για να δούμε τι σημαίνει για την Επιτροπή μας χρειάστηκε να συνεργαστούμε ε, και ε, για τα θέματα της ανθρωπιστικής βοήθειας και των επιπτώσεων σε αυτή. Λοιπόν, για να κλείσω λίγο την συζήτηση γρήγορα. Η, η βασική αρχή είναι μια αρχή που θα πρέπει να γίνει δεκτή, σεβόμενη το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί να ασκηθεί μέσω μιας χρήσης στρατιωτικών μέσων, που δεν θα πρέπει να συγχαίεται με τον ρόλο των ανθρωπιστικών εμπλεκομένων εταίρων, γιατί πρέπει να κάνουμε τη διάκριση, γιατί αυτό θα είναι εις βάρος και θα οδηγεί στον τερματισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η πρόληψη θα πρέπει να είναι το κεντρικό σημείο της προσπάθειας, έτσι ώστε η, η να μην υπάρχει ανάγκη παρέμβασης. Η ευθύνη προστασίας μπορεί να προχωρήσει και μέσω διπλωματικών μέσων, όπως η δημιουργία τοπικών μέσων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρηστή διακυβέρνηση και ένα σύστημα ε, έγκαιρης προειδοποίησης. Τα αναγκαστικά μέτρα και οι κυρώσεις ε, και η διαμεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει. Η κοινωνία των πολιτών οι περιφερειακές ενώσεις κρατών και οι διεθνείς οργανισμοί καλούνται να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτήν την διαδικασία μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Η γνωμοδότηση την οποία θα συγγράψω εξ ονόματός σας θα εμένει σε αυτές τις ε, αρχές. Και θα δεχθώ τροπολογίες και στο υπάρχον κείμενο για να υπογραμμιστεί ο ρόλος της πρόληψης και στον τομέα της, του δικαιώματος και του καθήκοντος προστασίας παράλληλα με τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αφρικανική Ένωση ήταν πρωτοπόρος στην αρχή σύμφωνα με την οποία η διεθνής κοινότητα οφείλει να παρεμβαίνει στην περίπτωση όπου υπάρχουν μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος αποτυγχάνει να τις αντιμετωπίσει. Τώρα, το δικαίωμα της προστασίας και οι μελλοντικέ εξελίξεις θα πρέπει να συμβαδίζει με την διεθνώς ισχύουσα ανθρωπιστική τάξη και δίκαιο. Αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία εκ νέου για τη βοήθειά της, για το κείμενο, το πρώτο που έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέρενς, έχετε τον λόγο. Να ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάικολ, ο οποίος επιτέλους θα κατάφερε να έρθει εδώ και για το πώς μας παρουσίασε το R2P, την ευθύνη προστασίας. Ε, κατά την απόψη μου, το Responsibility to Protect είναι το καλύτερο έγγραφο που μπορούσαμε να προτείνουμε στο πλαίσιο των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της ε, φτώχειας και της ανασφαλείας. Είναι εξαιρετικό έγγραφο, αλλά δυστυχώς αυτό το έγγραφο δεν κατάφερε να μετατρέψει σε κανόνες τις έννοιες που περιλαμβάνει το Responsibility to Protect. Επιπλέον αυτή η σύσταση χρησιμοποιείται ως αναφορά. Αυτή η αναφορά αρχίζει να συμπεριλαμβάνεται στα ψηφίσματα των Ομονεθνών ειδικά στη Λιβύη, όπου έγινε αναφορά για τις έννοιες που συνέταξαν οι συντάκτες του Responsibility to Protect. Είναι καταπληκτικό αυτό το εγγραφό διότι λέει τα πράγματα πάρα πολύ καθαρά και ειδικότερα κάνοντας διάκριση μεταξύ άμεσων και υποκείμενων ενιών και ε, αιτιών διανέξεων. Δηλαδή, σημεία ελάσσονες σημασία που μπορεί ωστόσο να ξεχυλήσουν το ποτήρι και να οδηγήσουν σε σημαντικά προβλήματα. Αλλά επιμένει κυρίως στις κρυφές αιτίε ε, όπως είναι η φτώχεια. Η φτώχεια συνά είναι συνώνυμο της απουσίας διακυβέρνησης σε εθνική ή τοπική κλίμακα. Είναι αλληλοσυνδεόμενοι αυτοί οι δύο παράγοντες. Είναι ένας πραγματικός φαύλος κύκλος. Το ζήτημα είναι να δούμε πώς μπορεί να κόψει κανείς, να σπάσει αυτό το φαύλο κύκλο. Ένα κράτος με ελάχιστους πόρους ε, χωρίς οικονομικές δραστηριότητες, χωρίς συνεπώς φορολογία, δηλαδή με κενό προϋπολογισμό, δεν μπορεί να επιτελέσει τις ε, λειτουργίες του, δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια για τους πολίτες του. Εδώ δηλαδή τίθεται το ζήτημα πρωτίστως των ερωτημάτων αυτών που αντιμετωπίζει ως θέματα το responsibility Το responsibility to protect και όλο το φάσμα παρέμβασής της μπορεί να εφαρμοστεί στις σημερινές διενέξεις στο Συρία, στο Σουδάν, στο Κονγκό, στη Τσετσενία, στα Δυτικά Βαλκάνια και κυρίως στο Μάλι. Όσον αφορά το Μάλι, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Δεν θέλω να είναι μετριοπαθής η στάση της Επιτροπής μας επί αυτού του θέματος. Αν υπάρχει μία επιτροπή που πολιτικά θα μπορούσε να συμβάλλει στην εξέβρεση λύσεων βάσει των διδαγμάτων του Responsibility to Protect, αυτή είναι η Επιτροπή Ανάπτυξης. Δεν πρέπει εμείς να είμαστε πίσω από τις υπόλοιπε επιτροπές. Πρέπει να είμαστε στο προπύργιο. Πρέπει να συμμετέχουμε σε όλες τις συζητήσεις ισότιμα με τις άλλες επιτροπές, διότι εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει να προτείνουμε λύσεις αυτή τη στιγμή η στρατιωτική λύση έχει φτάσει στα ωριά της. Μην με παρεξηγείτε, είμαι υπέρ της γαλλικής παρέμβασης στο Μάλι. Είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατάφερε και που γνωρίζει το έδαφος που κατάφερε να ανακόψει, να ανασχέσει την πορεία των τρομοκρατών που ήταν έτοιμοι να καταλάβουν τον Παμάκο. Όλοι γνωρίζουν ότι σε αυτή την περίπτωση τα στρατιωτικά μέσα δεν είναι ποτέ οι τελευταίοι ε, στην, ε, στους επεμβαίνοντας. Η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να δει πώς θα μπορέσει να ε, κάνει τους τρομοκράτες να εγκαταλείψουν αυτά τα έφορα εδάφη του Μάλι θα πρέπει επίση όμω, και ευχαριστώ τον Μάικλ που το ανέφερε στη συζήτηση, θα πρέπει να καταλήξουμε σε κατάλληλα συμπεράσματα όσον αφορά το πώ θα οργανώσουμε τι εργασίε μα. Ευχαριστώ. Καθώ δεν ήσασταν ούτε ο ένα ούτε ο άλλο στην έναρξη τη σημερινή μα συνεδρίαση, θα, θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι ξεκίνησα μιλώντα για το Μάλι. Και θα ήθελα να σα πω ότι δυστυχώ ε, ήταν απαραίτητη η παρέμβαση, αλλά δεν μπορεί από μόνη τη να αρκέσει ότι πράγματι η Επιτροπή Ανάπτυξης έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη φάση μετά την παρέμβαση. Θα σας στείλω, ε, σας έχω στείλει μάλλον ήδη ένα αντίγραφο της δήλωσής μου. Δίνω το λόγο τώρα στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, κυρία Κριστίν Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζουμε και θερμά το γεγονός ότι στρέφει την προσοχή στην ευθύνη να προστατεύσει το Ευρωκοινοβούλιο στο σχέδιο γνωμοδότησης αλλά και στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στην οποία συνεισφέρει. Η υποχρέωση προστασίας είναι ένα από τα θέματα κλειδιά στην δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ για, στα θέματα ασφάλειας. Είναι ένα θέμα όπου με συνέπεια προσπαθούμε να προαγάγουμε αυτό, αυτή την προσέγγιση και την παγίωση, την εμπέδωση αυτής της προσέγγισης αλλά και την εφαρμογή της. Και συμμετέχουμε ενεργά στην ετήσια συζήτηση και αυτό έρχεται σε μια πολύ καλή χρονική στιγμή ως πρωτοβουλία. Να συνεισφέρουμε σε μια συζήτηση που θα γίνει κανονικά τον Ιούνιο στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πραγματικά στην πρόληψη θα είναι επικέντρωση. Πρόληψη. Ε, σε αυτό επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΟΗΕ. Όχι μόνο κατά το προηγούμενο έτος, αλλά από τότε που το ψήφισμα του, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υιοθετήθηκε και η συζήτηση διεξήχθη υπό το πρίσμα αυτό και για την πρόληψη επίσης όσον αφορά και τη συνεισφορά της ε, διεθνούς κοινότητας για τη διαμεσολάβηση και τη δυνατότητα αυτής της δραστηριοποίησης που αναφέρθηκε στην γνωμοδότηση αλλά και το δυναμικό που μπορεί μακροπρόθεσμα να δομηθεί ώστε να προστατεύονται οι πληθυσμοί από τέτοιες ομότητες. Σίγουρα θα εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή, θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο, στη γνωμοδότηση και σε σχέση και με το περιεχόμενο του ψηφίσματος. Ένα άλλο θέμα, και θα είμαι σύντομη, είναι ότι προφανώς επίσης καλωσορίζουμε και πλήρως ημεριζόμεθα το, τις απόψεις για το θέμα για την ανάγκη να προστατεύεται η ανθρωπιστική δράση και δραστηριοποίηση και επίσης η αναφορά σας στο πλαίσιο του ε, διεθνού, ε, διεθνούς ε, νομοθετικού πλαισίου ως σημείο αναφοράς. Ευχαριστώ. Merci. Merci Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Κάσμαν για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκέρενς. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας, Charles. Και πραγματικά πρέπει να υπενθυμηθεί εδώ ότι δεν υπάρχει δεσμευτική ισχύς σε σχέση με το δικαίωμα προστασίας. Είναι ένα σημείο αναφορά αυτό το έγγραφο. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ότι το έγγραφο αυτό συνεπώς ε, με συνέπεια θα υπομνηματίζεται και θα αναφέρεται ως σημείο αναφοράς. Δική μας δουλειά είναι ακριβώς να επικεντρώσουμε και να δώσουμε προσανατολισμού σε εκείνους που θα δραστηριοποιούνται στα αναγκαία στοιχεία που θα εμπεριέχει αυτό το έγγραφο. Και σίγουρα είναι σωστό, υπάρχει υποχρέωση να αντιμετωπιστούν τα αίτια της φτώχειας, της κακής ή απουσίας διακυβέρνησης, της απουσίας συλλογής φόρων και να υπάρχει η αναφορά σε σχέση με τις δυτικές χώρες όταν υπάρχει τέτοια απουσία συλλογής ε, ε, κονδυλίων από πλευράς φόρων και της ε, αποδυνάμωσης των κυβερνήσεων και των καθεστώτων των αναπτυσσομένων χωρών. Και για το πλαίσιο αναφοράς για το δυναμικό ε, όσον αφορά την ε, ικανότητα προστασίας και πάλι αυτό πρέπει να είναι ένα σημείο αναφοράς. Και πάλι να μην αγνοήσουμε τις εξελίξεις. Είδαμε και μία 10% περικοπή των κονδυλίων που προτείνεται από τον πρόεδρο Φαν Ρόμπα και, άλλων, ε, και από άλλους. Είναι φρικαλές οι συνέπειες μιας τέτοιας περικοπής. Θέλω να ολοκληρώσω. Το δικαίωμα προστασίας πρέπει στην εφαρμογή να περιορίζεται στα τέσσερα εγκλήματα που προανάφερα πιο πριν ως πυλώνες και πρέπει σαφώς να καθοριστεί ένα πλαίσιο ώστε να διασφαλίζεται η χρήση μέσα σε ένα συνεπές και αποτελεσματικό πλαίσιο η αποτυχία σε σχέση με την ε, Συρία, η αναφορά στο, στη Λιβύη, η αναφορά στο Μάλι, όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη για να κατανοήσουμε πώς και πότε πολίτες, ε, πληθυσμοί πρέπει να προστατεύονται αν όχι από την ίδια τη χώρα τους, τότε από την διεθνή κοινότητα. Και τέλος ε, και από τις στάχτες και την καταστροφή που είδαμε στην Ρουάντα, αυτό θα πρέπει να αναδύεται και να θυμόμαστε ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να επιτραπεί να επαναληφθεί ποτέ ξανά. Και αυτό συνέβη επειδή σταυρώσαμε τα χέρια και το αφήσαμε να συμβεί. Και κάποιοι κέρδισαν κιόλα επειδή άλλοι δεν έκαναν καθόλου ή οι ίδιοι δεν έκαναν τίποτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Alors... Euh, λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι έχετε μέχρι την 30η Ιανουαρίου, 12 το μεσημέρι, για να υποβάλλετε ε, γνωμοδοτήσεις για τροπολογίες για την γνωμοδότηση του κ. Κάσπαν και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα 18 Φεβρουαρίου. Αν διακόπτεται τώρα η συνεδρίμασή μας, θα συνεχίσουμε αύριο στις 9 με τους συντονιστές, 10 η ώρα για τα μέλη. Καλό σας βράδυ. Υπότιτλοι